Ladies and gentlemen, good morning. Um, I know we've got... Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Ξέρω ότι έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ψηφοφοριών και μια μακρά ημερήσια διάταξη και με περίπλοκα θέματα για να συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Ε, κατόπιν τούτου και λόγω αυτών που συνέβησαν την Κυριακή θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας ε, με ένα λεπτό συγγύης προς ε, τη, μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκυριακό και για να σκεφτούμε όλοι μαζί την Ευρώπη. sure we all Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τα βαθιά μας ε, και ουσιαστικά μας ε, συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των ε, θυμάτων. Το πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξη είναι το θέμα των, των μπορείου και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Πρώτο θέμα λοιπόν η τροπολογίες 3 και 42 που είναι ταυτόσιμες υπέρ παρακαλώ κατά έλεγχος ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην τροπολογία 3 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπαρχών 3, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω πέρασε. Η 44 υπέρ, κατά, αποχές πέρασε. Η 4 και η 5 υπέρ, κατά, και η 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 5. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, καταπίπτει. Μισό λεπτό. Η τροπολογία υπαριθμών 5 παρακαλώ. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. καταπίπτη. Η 49 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει, η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 59 υπέρ, κατά αποχές καταπίπτει, η υπερθμόν 8 υπέρ κατά αποχές ε, καταπίπτει, η 60 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 9 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 61 είναι μια γλωσσική τροπολογία υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα που προβλέπει να προσθεθεί ή να υπάρχει ε, ορισμός τουλάχιστον 100.000 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο δεύτερο τμήμα, τροπολογία υπαριθμών 63 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 63. Συμβαστική δέλτα. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 15 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική ή e υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 υπέρ κατά Μισό η συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 79 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 86 υπέρ, όχι, η 87 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 90 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Η 90 απορρίπτεται, 91 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 92 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, ε, 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 96 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1-2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. Η 104 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά τροπολογία συμβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, 35 και 36 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται η 37 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 39 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται ή 40 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε για τη γνωμοδότηση στο σύνολό της, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζατε όλοι. That's passed. Thank you to everybody who worked extremely hard on that. Ευχαριστούμε όλους και παρότι δεν πέρασε ε, ομόφωνα. Υπήρξε αρκετά μεγάλη συμφωνία για πολλά ε, κομμάτια και τμήματα της ε, έκθεσης αυτής. Παρακαλώ. Επόμενο σημείο. Εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση. Σύσταση από δεύτερη ανάγνωση. Από ό,τι φαίνεται θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Two more to vote. Ψήφισαν όλοι. Όχι. So that's 33 to 1. Congratulations. 33 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Ευχαριστώ. Ε, συγχαρητήρια, Ανδρέας. Περνάμε επομένως τώρα. Α, όχι, αυτό τώρα θα πάει στην Ολομέλεια. Συγχαρητήρια. Επόμενο θέμα γνωμοδότηση για την έναρξη μέρους διαλόγου το 2017 είναι η έκθεση της κυρίας Γιάκων Σάρη τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ηλεκτρονική επαλήθευση αν θέλετε, ναι. Καταπίπτει. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, και ε, ψηφοφορία επί του συνόλου της γνωμοδοτήσεως. Σας ευχαριστώ και επομένως εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία ευχαριστούμε Λίσα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Ε, σας παρακαλώ να ηρεμήσουμε και να φτάσουμε στην αναθεώρηση της οδηγίας για τον έλεγχο των ε, όπλων. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Βίκη Φόρτ. Συζητάμε σήμερα για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Να σας πω ότι όπως ξέρετε έχουν υποβληθεί ε, πολλές τροπολογίες. 903 συγκεκριμένα μαζί με τις επιτροπές ε, ΛΥΜΠΕ. Η συγγήτρια είναι λοιπόν η πρόεδρός μας κυρία Φόρντ και επομένως θα της δώσω άμεσα το λόγο έτσι ώστε να παρουσιάσει ε, τα στοιχεία της και μετά θα, συνεχίσουμε με τους υπολείπους, ε, δηλαδή τους κοιόδης εισηγητές, ε, την Επιτροπή τα λοιπά. Παρακαλώ κυρία Φόρντ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι πολλοί θα παρακολουθούν και εκτός από την αίθουσά μας αυτή τη συνεδρίαση ένας πολύ μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και έπαφων εκτός κοινοβουλίου δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Να υπενθυμίσω λοιπόν σε όλους γιατί εξετάζουμε αυτά και τα προσεγγίζουμε Υπάρχουν ε, προφανώς εδώ και 25 χρόνια κοινά νομοθετικά ε, εγχειρήματα και μετά από τις επιθέσεις των Παρισίων ήταν σαφές ότι υπήρχαν κενά στη νομοθεσία όσον αφορά τη, της, ε, τη χρήση και την κατοχή ε, όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις, νέες προτάσεις για να ρυθμιστεί αυτό ο τομέα Και είναι απόλυτα θεμητό και σωστό να επανεξεταστεί νομοθεσία και να κλείσουν τα κενά. Και στο πρώτο σχέδιο του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφές ότι υπήρχε ισχνή πενιχρή διατύπωση και υπήρχαν πολλές ε, χωρίς πρόθεση ε, αρνητικές επιπτώσεις. Και θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω συνολικά τους συναδέφους για τις πολλές διαφορετικές τροπολογίες τους, αρκετές εκατοντάδες από την Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα να επεξηγήσω για τον τρόπο που θα συνιστούσα να την ε, αποδοχή, την δομή και αποδοχή των συμβιβασμών. Προτείνω λοιπόν έτσι να κατατεθούν και να εγκριθούν. Θέλω να ευχαριστήσω τις διαφορετικές πολιτικές ομάδες που ήδη κατέθεσαν γραπτές ε, προτάσεις και σχόλια σε αυτούς τους συμβιβασμούς. Για το πρώτο θέμα, για τα πυροβόλα όπλα, υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία για το ότι πραγματικά αυτά τα όπλα θα πρέπει να θεωρούνται ως ε, ε, επικίνδυνα και θα πρέπει να πολλούνται μόνο σε άτομα που έχουν άδεια να τα φέρουν. Δεύτερον, πρέπει να βεβαιώσουμε ότι άτομα που δημιουργούν κίνδυνο για τον ίδιο τον εαυτό τους ή άλλους δεν θα πρέπει να την χάνουν αδειοδότησης μέσω του νόμου και γι' αυτό θα έπρεπε κάθε χώρα να έχει ένα σύστημα το οποίο θα ε, έχει θεσπιστεί, θα έχει εγκριθεί ώστε να αποφασίζει η νομοθεσία της χώρας αυτής αν θα δίνεται η άδεια ή όχι ένα μόνιμο σύστημα δηλαδή ή ένα σε τακτές, ε, για τακτά διαστήματα ε, σύστημα που θα ρυθμίζει αυτά τα θέματα και θα πρέπει μετά να δούμε αν αυτό εγκρινόμενο μπορεί να προχωρήσει στη ρύθμιση αυτή. Ένα άτομο αν δεν τύχει αδειοδότησης ε, για τέτοιου είδου όπλα σε μια χώρα, οι αρχές των άλλων κρατών θα έπρεπε να μπορούν να γνωρίζουν αυτό το γεγονός ότι έτυχε άρνησης ε, όταν περνά σε μια άλλη χώρα πρέπει να είναι πολύ εύκολο για τις αρχές αυτής της χώρας να γνωρίζει αυτή την αρνητική έκβαση αυτής της αίτηση. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη ροή πληροφοριών είτε μέσω αυτόματων συστημάτων ε, ειδοποίησης είτε μέσω κομβικών σημείων επικοινωνίας ώστε να είναι το ευρωπαϊκό σύστημα πιο αποτελεσματικό. Υπάρχει και μεγάλη συνένεση για να υπάρξουν νέες απαιτήσεις για την ασφαλή αποθήκευση. Με όλες ε, τις χώρες όπου έχουν γίνει συζητήσεις υπάρχει αυτή η πρόθεση, αυτή η ρύθμιση και υπάρχει και μεγάλη υποστήριξη και από το Ευρωκοινοβούλιο προτείνουμε μια νέα διατύπωση όσον αφορά την τυποποίηση, τον χαρακτηρισμό αυτών είτε πρόκειται για τέτοιου είδους όπλα είτε για εξαρτήματα τα οποία μπορούν ίσως να απολυθούν ξεχωριστά για τέτοιου είδους όπλα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία που θα εγκρίνουμε θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και λειτουργική ώστε να είναι εύκολο να ε, σημαδευτούν και να χαρακτηριστούν με αυτόν τον τρόπο τέτοιου είδους όπλα και εξαρτήματα και για τον ρόλο των οπλοεμπόρων ε, ε, θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα είναι μόνο τότε επιτρεπτό όταν θα έχουν καταχωρηθεί, θα έχει εξεταστεί η ταυτότητα των ετούντων και όσον αφορά και τη διαχείριση ε, ιστορικών συλλογών ή όπλων. Προτείνουμε πρώτα να ρυθμίσουμε και να δούμε αν αυτό θα τεθεί εκτός πλαισίου, αυτή τη στιγμή εξαιρούνται και θα πρέπει να ψηφίσουμε αν αυτή η εξαίρεση θα συνεχίσει να υφίσταται ή όχι. Και αν αυτό καταπέσει τότε θα ψηφίσουμε για το αν ή όχι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνουν τέτοιες άδειες σε επίπεδο κρατών μελών. Θα υπάρχει λοιπόν διτή δυνατότητα να ρυθμιστεί αυτό. Η εξαίρεση κράτους μέλους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτού του είδους τα όπλα να μπορούν να αποθηκεύονται με ασφάλεια σε σχέση με την νομοθεσία ως έχει, έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν εξαιρέσεις στα κράτη-μέλη και είναι πάρα πολύ σημαντικές για οργανώσεις όπως ε, ε, βαλιστικούς πραγματογνώμονες, ε, κατασκευαστές και προτείνουμε τα κράτη-μέλη να μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν τέτοιου είδους εξαιρέσεις για την κατηγορία Α για την εξαίρεση αυτή στο αντίστοιχο άρθρο έχουμε αποσαφηνίσει με τη διατύπωση το τι πρέπει να γίνεται για την εθνική άμυνα είναι ζωτική σημασίας τα κράτη-μέλη και οι στρατιωτικές τους δράσεις και τα αμυντικά θέματα ε, των οποίων επιλαμβάνονται να μην ε, υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις από τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Πρόκειται και για ένα πολύ τεχνικού χαρακτήρα θέμα και πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι ένα όπλο μόνο τότε θα μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ε, αδρανοποιημένο αν δεν μπορεί να μετατραπεί με τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση του να μπορεί να, να, να χρησιμοποιηθεί το όπλο αυτό ως ε, πυροβόλο όπλο. Γι' αυτό θα πρέπει με αυτή την αδρανοποίηση, εξουδετερώση, μόνιμα να εξουδετερωθεί. Το πρώτο σχέδιο για την ε, εξουδετερώση το οποίο εγκρίθηκε από τις τεχνικές ομάδες των κρατών μελών τον Νοέμβριο 2015 προκάλεσε πολλές πολλά θέματα ε, εφαρμοστικότητας, εφαρμογής που έπρεπε να εξεταστούν και λόγω απουσίας ε, σαφούς διατύπωσης και γι' αυτό στα παραρτήματα αυτό που προτείνουμε είναι να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά τις κανονιστικές και αριθμιστικές ε, διατάξεις. Αν μπορέσει με το τριμερή διάλογο αυτό να επιτευχθεί, σε σχέση με την έγκριση τροποποιήσεων αυτού του κανονισμού αν έγκαιρα θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τότε αυτό μπορεί να ρυθμίσει το θέμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Πρέπει όμως αυτό να αποσαφινιστεί οπωσδήποτε διότι υπάρχουν πολλά τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα με αυτές ε, τις ρυθμίσεις και αρκετά από αυτά έχουν ε, και επιπτώσεις όσον αφορά την θέματα ασφάλειας. Έχουμε από την άλλη πλευρά επίσης ε, προβλέψει και νέες προτάσεις όσον αφορά τις υφιστάμενες διατάξεις εξουδετέρωσης και όπου υπάρχουν τέτοιες ε, προδιαγραφές από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζονται για τις κατηγορίες Α και Β και αυτό είναι μάλλον το πιο επίμαχο ζήτημα αυτής της ρύθμισης και γι' αυτό η σύστασή μου είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της δημοκρατίας εδώ. Ένας βουλευτής πρέπει να έχει την δυνατότητα αναρρύθμιση να εγκρίνει, να απορρίψει τις διατάξεις για τα όπλα αυτά όσον αφορά την προσθήκη ή την ένταξη κάποιου όπλου στον ε, πίνακα απαγορεύσεων. Υπάρχει εδώ ε, έντονα η αίσθηση ότι το άρθρο Α7 της Επιτροπής ε, δεν είναι λειτουργικό και δεν μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να δημιουργήσει μια κατάλληλη μέθοδο για, τον, για τη ρύθμιση του αν κάτι θα απαγορεύεται ή όχι. Γι' αυτό για το Β7 υπάρχουν και αρκετές ρυθμίσεις ε, που διατυπώθηκαν για να προσθεθούν και άλλα τέτοια αντικείμενα στον ε, κατάλογο αυτό. Κάποια από αυτά προέρχονται και από το ίδιο το Συμβούλιο. Η πρότασή μου είναι να ψηφίσουμε αυτά και να ρυθμίσουμε έτσι το ζήτημα. Υπάρχουν ανησυχίες από κάποια κράτη-μέλη για το θέμα των αυτόματων πυροβόλων όπλων που έχουν μετατραπεί σε ήμια αυτόματα πυροβόλα όπλα. Και εδώ υπάρχουν και θέματα ασφάλειας ε, και ανησυχίες. Αν μήπως αυτά όταν απαγορευτούν δεν παραδοθούν στις αρχές αλλά με παράνομο τρόπο συνεχίσει να υφίσταται κατοχή αυτών των όπλων από ιδιώτες. Πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και να το αντιμετωπίσουμε. Αν η πρώτη εναλλακτική λύση θα ήταν να απαγορευτούν ή αν από την άλλη πλευρά αποφασίσουμε ότι μπορούν να διατηρηθούν τότε υπάρχει πρόταση να ε, οι, διατάξεις για τη μετατροπή να διασφαλίζουν ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα αυτή η μετατροπή αυτών των όπλων. Και τελευταία παρατήρηση για την πρόταση του Συμβουλίου από την προηγούμενη εβδομάδα που έχει και κάποιες κατηγορίες ε, όπλων ε, της κατηγορίας Α ανάλογα με το δυναμικό πυρός που έχουν, τη δύναμη πυρός που έχουν θα έπρεπε λοιπόν νομίζω να ε, εξεταστεί το θέμα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Γνωρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε καταθέσει συμβαστικές τροπολογίες για τις αιτιολογικές σκέψεις, διότι αυτές πρέπει να αντανακλούν αυτά τα οποία θα συνεπάγεται το έργο μας ε, για τα επιμέρους άρθρα. Εστιαζόμαστε στα άρθρα, πρέπει να εστιαστούμε επί των άρθρων πρώτα και μετά να επανέλθουμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στους, στους ε, ε, σκιώδη, Αντα Μαρία Κοράτσα Μπίλντ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Βίκη, την εισηγήτρια. Ήταν ε, πολύ καλό που δούλεψα μαζί σου, το χάρηκα και ε, με πολλά σημαντικά στοιχεία έχεις παρουσιάσει. Να υπενθυμίσω λίγο το πλαίσιο. Είχαμε μια αρχική πρόταση από την Κομισιόν, η οποία ούτε ισορροπημένη ήταν, ούτε σωστή σωστή. Γι' αυτό λοιπόν ε, ζητήσαμε να την τροποποιήσουμε. Δείξαμε ότι ε, το Κοινοβούλιο πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση με πιο εστιασμένη, ε, με μεγαλύτερη συγγνώμη εστίαση στην ασφάλεια χωρίς να καταστέλλονται οι ελευθερίες ε, των ε, ανθρώπων. Βεβαίως πρέπει να εξυγχρονιστεί ε, η νομοθεσία και αναφέρθηκε ήδη στην καταχώρηση, στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής ε, νόμου, ταυτοποίηση, δυνατότητα ταυτοποίηση ε, των όπλων, ε, την ίχνηλασιμότητα, την σήμανση η οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά. Ταυτόχρονα με τους συμβιβασμούς προσπαθούμε να μην αυξήσουμε το διοικητικό ε, και γραφειοκρατικό άχθος για αυτούς ε, που νομίμως κατέχουν ε, όπλα. Επίσης όμως έχουμε αναφερθεί και στην ασφαλή αποθήκευση, πράγμα που δεν αναφερόταν στην αρχή. Είναι σημαντικό να έχουμε και ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για τις δοκιμές ε, και επομένως ε, ε, ένα πλαίσιο δηλαδή που να μην τροποποιεί αυτούς που ήδη έχουν ένα ικανό πλαίσιο αλλά να αυξηθεί η προστασία για αυτούς που δεν έχουν. Η πενταετία που ανέφερες επίσης είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Δεν θέλουμε βεβαίως να δημιουργήσουμε και πρόβλημα σε όσους ζουν στην Ήπεθρο και που νομίμως μπορούν να αγοράσουν και να συμμετέχουν να έχουν στην κατοχή τους ε, όπλα. Επίσης όσον αφορά τους εθελοντές, όσον αφορά ε, τους ε, στρατολογούμενους κλπ. για λόγους άμυνας οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα για πυροβόλα όπλα. Όσον αφορά τώρα ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω η παράγραφος 1C νομίζω ότι θα πρέπει να διαγραφεί διότι θα πρέπει κατά τη δική μου άποψη να αποτελεί απόφαση απόφαση των κρατών μελών. Όσον αφορά την ε, ε, ασφαλή αποθήκευση, νομίζω ότι δεν πρέπει να αναφερθεί εκεί το θέμα των μεταφορών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όσοι έχουν ε, ασφαλώς αποθηκευμένα όπλα να καλύπτονται κτλ. Εκεί μετά θα διαγράψουμε την συνέχεια μέχρι, μέχρι την μεταφορά και να συνεχίσουμε μετά την ε, με την υπόλοιπη φράση είναι το ένα d και όχι το ένα c Έκανα λάθος λέει η ομιλήτρια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της... η χειρονακτική χρήση, η αναγόμωση του ε, όπλου και νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να μείνουν απλά και ε, σαφή. Ε, όσον αφορά τα κύρια συστατικά, ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει στο σώμα της ε, του νομοθετήματος να αναφερθούμε σε αυτό. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο για τα πυροβόλα όπλα που το καλύπτει. Τελευταίο που θέλω να πω είναι το θέμα των παραρτημάτων. Ήδη Βίκη το ανέφερες ότι δεν θα πρέπει να ε, να απαγορεύουν την κατηγορία των ημιαυτομάτων ε, όπλων. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να προσθέσουμε την κατηγορία Α7 ε, γιατί τώρα το να ρυθμίσουμε τέτοια στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καθόλου καλό κατά την άποψή μου. Βελινετική και τέτοια πράγματα. Ε, ε, όσον αφορά τώρα τα μουσεία και τα συλλεκτικά όπλα, συλλογέ κτλ. θα πρέπει το κείμενο να παραμείνει ε, απαράλλακτο και δηλαδή να παραμείνει το κείμενο τη Κομισιόν και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε την καλή συνεργασία και θα έχουμε ένα καλό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ανα Μαρία Κοράτσα Μπίλτε, ο Σέρτζο Κομφεράτη για του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω την Βίκη για τη δουλειά που έκανε και για τις ε, τροπολογίες που ήταν πάρα πολλές γιατί το θέμα είναι πολύ περίπλοκο ε, υπάρχουν και διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, άρα δηλαδή ε, έπρεπε να βρεθούν κάποια σημεία συγκλήσης, κάτι το οποίο αν ξεκινάει κανείς από μεγάλη απόσταση δεν είναι εύκολο να υπάρξει σύγκληση. Εμείς ε, ως ομάδα ε, χθες το βράδυ ε, παρουσιάσαμε τη στάση μας στην εισηγήτρια και στους άλλους και εισηγητές. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά εδώ να αναφέρω κάποια θέματα τα οποία έχουν σχέση περισσότερο με τη μέθοδο. Διότι στο κείμενο το οποίο ή στα κείμενα που μας έδωσε η δίκη. Υπήρξαν κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικέ λύσεις. Υπάρχει μία μέθοδος εργασίας, η οποία μπορεί αρχικά βέβαια να είναι αποτελεσματική, μετά όμως μπορεί και να ξεπεριστεί. Άρα δηλαδή μας, μας ενδιαφέρει να αναζητήσουμε συγκλίνουσες διατυπώσεις, οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Και αν δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει παρόλα αυτά να υπάρχει μία αναλλακτική λύση η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, μεθόδου ε, και κάποια στιγμή θα πρέπει βέβαια να καταλήξουμε ε, πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία. Καλύτερα να εκφράζει κανείς ε, την ε, διαφωνία του, ε, γιατί δεν είναι εύκολο να υπάρχουν λακτικές λύσεις οι οποίες είναι και δυσνόητες. Εγώ νομίζω ότι πάντα όσον αφορά τη μέθοδο υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, να φανταστεί κανείς ότι για πάρα πολλές σημαστικές προτάσεις που κατέθεσε η συγγήτρια, πριν φτάσουμε καν στην πληροφορία, ε, διαγράφεται μια συγκεκριμένη παράγραφο Μα δεν γίνεται αυτό. Για να φτάσει κανεί σε μια σημαντική λύση πρέπει να υπάρχει μια σύνθεση πολιτικών στάσεων. Εάν εκ των προτέρων διαγράφει κανεί τα στοιχεία εκείνα τα οποία αφορούν στην πρόταση, ε, τι σύνθεση να γίνει. Προκύπτει κάτι λίγο διαφορετικό πράγμα. Ε, αποδοχή, αν θέλετε, τη ε, αρχική διατύπωση που μπορεί κάποιοι να συμφωνούν, αλλά ε, παρόλα αυτά αυτό δεν είναι αποδεκτό. Κατά την άποψή μου λοιπόν θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Κάτι άλλο. Όσον αφορά όλα αυτά, βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη φάση των εργασιών μας. Είναι και η τελική φάση. Επί των συμβαστικών προτάσεων θα ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα. θέματα τα οποία τα θεωρώ πιο ευαίσθητα και πιο σημαντικά από κάποια άλλα. Πρώτον, όσον αφορά την ανέωση της άδεια, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μια αρχική επαλήθευση της κατάστασης υγείας του ανθρώπου που έχει άδεια οπλοφορίας. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορεί να καταλήξει το όπλο στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν είναι σε φυσική και σωστή φυσική κατάσταση για να το χρησιμοποιεί είτε και είναι κάποιος ε, που το χρησιμοποιεί για αθλητισμό είτε για κυνήγι. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σίγουροι για τη φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Υπήρχε μια αρχική διατύπωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ δεν το ξαναείδα όμως μετά στις τροπολογίες. Ίσως πρέπει να επαναφέρουμε αυτή την διατύπωση ή εν πάση περιπτώσει να βρούμε κάποια λύση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξαποστάσεως πωλήσει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λείπει, εντάξει σωστό είναι το πνεύμα που διέπει όλη την τροπολογία, αλλά δεν γίνεται λόγος ε, για, την, ε, για τον έλεγχο που θα πρέπει να γίνεται σχετικά με την πώληση ενός όπλου. Δηλαδή να ελέγχουμε αυτός για τον, στον οποίο πρόκειται να απολυθεί πράγματι εκεί που λύθηκε, να ελέγχεται ο τελικός αποδέκτης. Και αυτό είναι σημαντικό, να προστατεύουμε τις εξαποστάσεως πωλήσει. Αυτό πρέπει κάπως να το δούμε. Όσον αφορά τα επιθετικά όπλα, νομίζω ότι εκεί πρέπει να εξαλειφθεί λιγάκι το θέμα των εφέδρων. Και θα πρέπει να βρούμε κάτι πιο καλό από αυτό που λέει το άρθρο 6. Πρέπει να λυθεί το θέμα των εφέδρων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εκεί να εξεταστεί το πρόβλημα. Στο 6. Καλύτερα στο 6 παρά στο άρθρο 2. Τώρα, για τα για τις συλλογές ε, στα μουσεία. Εντάξει, εκεί δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Το μουσείο πρέπει να ελέγχει τα εκτέματα και τις ε, συλλογές ε, και θα πρέπει να ελέγχει τον ενδεχόμενο μιας κατάλληλης χρήσης. Υπάρχει ένα εθνικό μητρό όπου καταγράφονται ε, τα όπλα ή θα πρέπει να υπάρχει, θα ήταν χρήσιμο αυτό σε αυτό το Εθνικό Μητρό. Ξέρετε, αυτό που δεν με πείθει είναι ότι αυτά που ισχύουν για τα μουσεία δεν πρέπει αυτόματα να ισχύουν και για τους συλλέκτες. Άλλο συλλέκτες, άλλο μουσεία. Οι συλλέκτες είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν και να διατηρήσουν τα όπλα αυτά στο σπίτι τους. Και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και αυτοί καλύπτουν τα κριτήρια που προβλέπονται για τα μουσεία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί μια κατάλληλη διατύπωση, ένας ορισμός τι σημαίνει συλλέκτης. Δεν αρκεί να λέμε ότι είναι φυσικό πρόσωπο. Δεν φτάνει αυτό. Φυσικά πρόσωπα είναι και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ε, συλλέγουν όπλα, αλλά συλλέγουν αν θέλετε και άλλα αντικείμενα. Τέλος, όσον αφορά τα παραρτήματα, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές προτάσεις. Ε, αυτά που προτείνει η Βίκη είναι σωστά, να μπουν στη συμβαστική πρόταση. Με περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε λιγάκι περαιτέρω τους ορισμούς και την κατηγορία Α6. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και μάλιστα θα το κάνουμε με την ίδια αφοσίωση και προσοχή που το κάναμε και για τα άλλα κεφάλαια. Βεβαίως έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία κάναμε μέχρι τώρα είναι ορμόμενα από θετικές ε, προσεγγίσεις και από μία έρευνα ε, που διεξήχθη. Ε, στην αρχή είχαμε πολλές αμφιβολίες. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με την ίδια αφοσίωση και με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Τσελεντσόβα, η κυρία Τσελεντσόβα από την Άντε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Βίκη Φόρντ για την ε, πολύ σκληρή δουλειά που έκανε. Δεν ήταν εύκολο αλλά καταφέρατε να ε, ε, να έχετε μαζί σας όλους όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα και τους απασχολεί το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθειά σας αυτή. Όπως γνωρίζουμε, την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε η Γενική Προσέγγιση από το Συμβούλιο. Η συζήτηση δεν ήταν εύκολη και πρέπει να πω ότι ε, το, η έκβαση δεν είναι καθόλου ε, τέλεια. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα βασικά στοιχεία, βασικά δηλαδή ε, όσον αφορά την ΑΛΤΕ. Από τον Νοέμβριο εμείς δεν ε, ε, συμφωνούμε με την διάταξη αυτή η οποία θα σήμαινε μαζική κατάσχεση όπλων από ε, το ευρύ κοινό. Αυτό κατά την άποψή μας θα πρέπει να αναφερθεί μονάχα και να αφορά μόνο τα ημιαυτόματα όπλα. Υπάρχει μια Ολλανδική πρόταση η οποία όμως επαναλαμβάνει την πρόταση της Κομισιόν και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάποιες δημοσιεύσεις των γενικών προσεγγίσεων ε, του ε, ε, Συμβουλίου μας έχει, είχε σαν αποτέλεσμα να κατακλειστούμε από επιστολές από τσέχους πολίτες εδώ, σε αυτή την Επιτροπή εμείς θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Πολλά κράτη συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας εδώ και χρόνια έχουν βρει καλή ισορροπία ανάμεσα στα θέματα ασφαλείας αφενός και τα δικαιώματα των κατόχων όπλων αφετέρου. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να προσπαθήσουμε ε, όχι να διαλύσουμε αυτήν την ισορροπία αλλά να την ενισχύσουμε περαιτέρω. Βίκη, υπάρχουν κάποιες προτάσεις στην, ε, ε, ή κάποιες εναλλακτικές στην πρότασή σου ε, και χαίρομαι που μας τις έχεις υποβάλει έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε σε σχέση με το τι θα πρέπει, ε, ε, η άποψή μας σχετικά με το τι θα πρέπει να επιτρέπεται και τι να απαγορεύεται θα πρέπει να είναι απολύτως ε, σαφή. Επίσης, για θέματα όπως είναι οι πωλήσει μέσω ίντερνετ ή εξ τα θέματα για τα μουσεία, τα θέματα για τους συλλέκτες, σε αυτά τα σημεία η άποψή σου με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Χαίρομαι που συνεργαστήκαμε και προσβλέπω στην επιπλέον επιπλέον συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σαρανσόβα. Δεν έχουμε ε, εξ ονόματος της ε, Γκουε τον υπεύθυνο εδώ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, ε, ο Πασκάλ Ντυρό για τους Φρασίνους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω εξ ονόματος της Γκουε γιατί δεν μου έχει δώσει τέτοια δικαιοδοσία. Και εγώ θα προσπαθήσω εν συντομία, γιατί βρισκόμαστε βέβαια ε, σε φάση μεγάλης και έντονης εργασίας ε, επί των συμβιβασμών, να ε, πω δύο λόγια, να ευχαριστήσω την Βίκη για μία ακόμα φορά, γιατί εδώ έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο, ένα από τα πιο ευαίσθητα της θητείας αυτής. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι για ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και σοβαρό δεν θα πρέπει ε, να ε, εκφράσουμε θέσεις ε, είτε υπερβολικές είτε ασύμβατες με την πραγματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη φάση δεν έχει καμία πρόταση ε, είτε από τη Βίκη Φόρντ είτε από κάποιον άλλο βουλευτή άνδρα ή γυναίκα, το κοινοβούλιο λέω, ε, με κανένα τρόπο δεν προσπάθησε με οποιαδήποτε πρόταση ε, να σπάσει την ισορροπία ή να απαγορεύσει την κατοχή πυροβόλων όπλων. Πουθενά δεν το είδα αυτό και θα ήθελα να διαβεβαιώσω όσους μας κατακλίζουν με mail ότι θα πρέπει να αγωνιζόμαστε με βάση την πραγματικότητα και όχι φαντάσματα. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε μια πρόταση από πλευρά της Κομισιόν ε, που ήταν μια ανεπαρκής πρόταση ε, όσον αφορά τους ορισμούς. Όλοι είπαμε εδώ ότι ε, η άρνηση των ε, ήμι αυτόματων όπλων με μόνο κριτήριο την ομοιότητά τους με τα αυτόματα όπλα δεν ήταν κάτι θετικό, δεν ήταν κάτι λογικό και το Κοινοβούλιο λοιπόν το τόνισε αυτό, είπε δεν είναι σοβαρό κριτήριο αυτό που μας υποβάλλεται, θα πρέπει να υποβληθούν πιο αντικειμενικά κριτήρια και σιγά σιγά τα καταφέρνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ευχαριστώ Βίκη για την εργασία που έκανες. Ε, πολύ ε, σύντομα γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, ε, παρατηρήσεις των πρασίνων ε, έγιναν δεκτές από την εισηγήτρια. Επομένως εγώ θα αναφερθώ πιο πολύ σε λεπτομέρειες, ε, ας πούμε να δούμε ποια, σε ποια σημεία μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις, δεν θα ζητήσουμε να καθορίσει η Ευρώπη τις ιατρικές εξετάσεις, αλλά η Ευρώπη μπορεί να ζητήσει να υπάρξουν ιατρικές εξετάσεις σε όλες τις χώρες οι οποίες θα γίνονται, οι εξετάσεις αυτές, ε, υπό την ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δηλαδή, ε, για την κατοχή πυροβόλου όπλου θα πρέπει να υπάρξει εκ των προτέρων ψυχιατρική και ιατρική ε, γνωμάτευση. Επίσης, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι ε, για ορισμένα πράγματα όσον αφορά ας πούμε ε, την, τον διαχωρισμό της φύλαξης. Μία, ένα σημείο για το ίδιο το όπλο, ένα σημείο για τα πυρομαχικά. Νομίζω ότι οι κάτοχοι των όπλων ήδη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια αποσαφήνιση. Όσον αφορά τις πωλήσει εξ Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται πραγματικός ε, και όχι πλασματικός έλεγχος. Ε, θα πρέπει να υπάρξει φυσικός, ε, φυσική επαφή και επαλήθευση έτσι ώστε να είναι επαληθεύσιμο το ποιος πραγματικά αγοράζει το όπλο, ποιος είναι πραγματικός αποδέκτης. Όσον αφορά την καταχώρηση των δεδομένων είμαι πεπισμένος ότι η καταχώρηση ε, που προτείνει η δίκη και που θα είναι προσβάσιμη από τις αρχές είναι κάτι καλό. Ε, τώρα η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ναι, δεν θέλω να δημιουργήσουμε καινούριε δομέ, αλλά νομίζω ότι μια πλατφόρμα μπορεί να είναι ένα σημείο ε, συνάντησης απόψεων και μπορεί να είναι κάτι χρήσιμο. Ε, μουσεία και συλλέκτες, ε, ο κύριος Σέζιο Κομφεράτη τα είπε πάρα πολύ ωραία συμφωνώ μαζί του. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα μουσεία που είναι ε, οργανισμοί ε, που ελέγχονται σαφώς, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, να τα ξεχωρίσουμε από τους ε, συλλέκτες. Όσον αφορά τις ταξινομήσεις έχουμε προχωρήσει. Πρόκειται για πολύ τεχνικό ζήτημα και δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι ναι, οι κατηγορίες α6, α7 ε, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί ε, κάποια λύση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε ε, με αυτό το θετικό πνεύμα συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντουράν για την EFDD, ο κύριος Ιβασκεβιτς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ εσάς για το έργο που επιτελέσατε. Αυτή η πρόταση είναι επίμαχο θέμα. Βλέπουμε ότι λείπει μια μελέτη επιπτώσεων σε σχέση με όλα αυτά. Και ίσως είναι αντιπαραγωγικό αυτό και πολλαπλά κιόλα. Προσπαθούμε βέβαια προφανώς να αποφύγουμε γεγονότα όπως τρομοκρατικές, ε, τρομοκρατικά πλήγματα. Όμως από την άλλη πλευρά για τα αθλήματα π.χ. για το κυνήγι που πρέπει κάποια πράγματα να ρυθμιστούν. Συμφωνώ για τα θέματα διαδότησης Όσον ε, επίσης ε, και με τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται. Εδώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι αυτόνομα στο ρόλο που θα ασκήσουν. Η πρώτη επιλογή, option one, πρώτη επιλογή φαίνεται να είναι καλύτερη. Πρέπει να γνωρίζουμε για τι πράγμα κάνουμε λόγο. Είτε θα είναι ψυχολογικές δοκιμασίες αυτές, είτε ε, ψυχικές, ε, ψυχιατρικές ε, ε, εξετάσεις. Διότι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την τρόπο μετακίνησης ε, που ε, συνεπάγεται πρόβλημα θα πρέπει να μην την χάνουν αδειοδότησης. Θα πρέπει να μπορέσουμε να μην ε, καταλήγουμε υπερβολικά συχνά σε τέτοιες καταστάσεις. Για το δεύτερο θέμα, για τη συμφωνία όσον αφορά την πρόταση της εισηγήτριας, θα έτεινα περισσότερο να υποστηρίξω την πρόταση της κυρίας Κάνασόβα. Επίσης συμφωνώ και με τα θέματα 3 και 4. Για την πρόταση για το 5 θα μπορούσαμε ουσιαστικά να συζητήσουμε το αρχικό, την αρχική διατύπωση για το άρθρο 9 παραστατιωτικές ομάδες και εδώ μάλλον θα πρέπει να πω ότι υπάρχει συμφωνία για την πρόταση της εισηγήτριας για τα παρατήματα, παράτημα 2 για το δεύτερο εδάφιο. Συμφωνούμε για το Β και το Γ, Β και Σ. Για το παράρτημα υπαριθμών 1, τμήμα 2, κατηγορίες Α, 6α. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοιχνευτεί και να, το, να, να εντοπιστεί ε, το παράτημα 1 για την ε, κατηγορία α, 6 και 6β τα πυροβόλα όπλα που απαγορεύονται, που χρησιμοποιούνται σε αθλήματα όπως ε, στην ε, ε, σκοπ, σκοποβολή. Ωστόσο αυτό δεν βλάπτει κανέναν. Ακούσαμε τι είπαν οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να διαπιστώσουν ότι υπάρχει οποιαδήποτε βλαπτική επίπτωση στη χρήση τέτοιων πυροβόλων σε σχέση με το 7α για παράδειγμα και την πρόταση να απαγορευτεί το εμπόριο τέτοιων όπλων. Ε, υπάρχει λοιπόν απόρριψη αυτής ε, της πρότασης, την απορρίπτουμε και το 7 πρέπει να ε, απαλληφθεί. Επίσης όσον αφορά τα όπλα διαμετρήματος 22 χιλιοστομέτρων στο Β, Πιστεύω ότι κάποιες ιδέες βλάπτουν πραγματικά το άθλημα της σκοποβολής στην Ευρώπη και δεν θα μπορέσουμε έτσι να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση και παρόμοιες ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ΕΝΕΦ e η κυρία Τροσίνσκι. Merci Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν αναφερθώ στο θέμα αυτό, ε, ξεκινήσαμε ε, με ενό λεπτού σιγή για τα θύματα του Ορλάντο και θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τη λύπη μου αλλά και το θυμό μου ε, μετά από τη νέα τρομοκρατική ενέργεια που γνώρισε η Γαλλία χτες και ε, να, ε, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τον θάνατο των δύο αστυνομικών ε, μετά από επίθεση με μαχαίρι από έναν τζιχαντιστή. Θα ήθελα να ζητήσω από την ε, κυρία Φόρντ τρία πράγματα. Να, αποσύρει τις, να αποσύρω τις τροπολογίες ε, της ομάδας μου επί τριών ε, συμβιβαστικών ε, τροπολογιών. Αλλά θα σας τα στείλω γραπτά με mail όσον αφορά τα ακουστικά όπλα ε, σήμανσης και, τις, και τα αντίγραφα. Τέσσερις τροπολογίες μάλλον ε, οι οποίες έχουν ε, μπει στο συμβιβασμό σας και που θέλω να αφαιρέσω από το συμβιβασμό αυτό. Επίσης, ε, όσον αφορά τα μουσεία και τους συλλέκτες, Επίσης θα ήθελα να αποσύρω την τροπολογία μας 616. Euh, Διότι δεν θα ήθελα ε, οι συλλέκτες να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της ε, οδηγίας. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με την αγγλική διερμηνία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την αγγλική διερμηνία, από ό,τι φαίνεται. Αποσύρετε τις τροπολογίες σας, αυτό είπατε. Γιατί άκουσα από τη διερμηνία ότι θέλετε να αφαιρέσετε. Όχι, δεν αποσύρω τις τροπολογίες μου. Αποσύρω τις τροπολογίες μου από τους συμβιβασμούς. Από, από εκεί τις αποσύρω. Αλλά θα σας τα πω θα σας κάνω ένα κατάλογο όλων των ε, τροπολογιών που επιθυμώ να αφαιρεθούν από τους συμβιβασμούς. Το καταλάβατε τώρα? Εντάξει, για να το απλουστεύσουμε ε, θα σας στείλω με mail όλες τις τροπολογίες τις οποίες η ομάδα μου επιθυμεί να αφαιρέσει από τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Πολύ ωραία. Λέει ο Πρόεδρος, τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, βουλευτές. Έχω 10 εγγεγραμμένους συναδέλφους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε και την κυρία Γιουροβά η οποία, την Επίτροπο η οποία θα έρθει. Ένα λεπτό ο καθένας ε, να προσπαθήσουμε όλοι λοιπόν να είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί. Μετά έχουμε και το Συμβούλιο έχουμε, ε, και έχουμε και την κυρία Φόρτ που θα πρέπει να πάρει το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχω κατανόηση για αυτό το θέμα των τροπολογιών και είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική συνένεση σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Έχουμε τώρα εκατοντάδες τροπολογίες. Θα πρέπει να επεξηγηθούν, να αποσαφινιστούν και θα ήθελα να γνωρίζουμε σαφώς ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι κοινοί κανόνες και απαιτήσει πρέπει να προβλέπονται από την άλλη πλευρά η πρόταση ως έχει μπορεί να πλήξει μια λάθος ομάδα ατόμων, λανθασμένη ομάδα. Έχουμε σκοπευτές και θύρευτες κυνηγούς στην Σουηδία και ενώσεις με μεγάλη παράδοση. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θέλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα αυτών των ατόμων και δεν θέλουμε να βρεθούν σε μειονεκτική μοίρα όσον αφορά την καταπολέμηση για παράδειγμα παράνομων όπλων και οπλισμού η μέχρι τούδε αντιμετώπιση είναι καλή και γι' αυτό πρέπει ξεχωριστά να δούμε τι θα γίνει για τέτοιου είδους κατηγορίες. Δεν είναι απόλυτα αναγκαίο οι κυνηγοί και οι σκοπευτές ε, να υποβάλλονται σε τέτοιου είδους ε, εξετάσεις ε, θα έπλητε με σοβαρό τρόπο αυτά τα άτομα αυτές τις ομάδες ανθρώπων. Ελπίζω ότι αφουγκράζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβει υπόψη αυτά. Δεν είναι δυνατόν αυτοί να επιβαρύνονται λοιπόν χωρίς λόγο οι κυνηγοί και σκοπεύουν. Σας ευχαριστώ. Έχετε, ε, υπάρχει αλληλεγγύη για αυτά τα θέματα. Δυστυχώς σε μια χώρα που η τρομοκρατία χαρακτήρισε την ε, ε, πρόσφατη ιστορία μας κατά τις πρόσφατες τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Γι' αυτό η νομοθεσία και ασφάλεια που υπάρχει στην Ισπανία για την ε, κατοχή όπλων είναι όχι μόνο υποδειγματική, αλλά επιπλέον για πολλά άτομα που έχουν νόμιμα όπλα, όπως κυνηγού, ε, σκοπευτές, ε, είναι πραγματικά δύσκολο να μπορέσει λόγω της μεγάλης πίεσης διοικητικής που υφίσταται να υφίσταται κάτι τέτοιο. σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά, αυτές οι προτάσεις εξετάσει ε, ε, εξετάστηκαν για χώρε οι οποίε δεν είχαν τέτοιου είδου ε, προβλήματα όπως στην Ισπανία. Τούτου λεχθέντος τώρα πρώτα θα ήθελα να πω στη συνέχεια ότι οι συμβιβασμοί της Βίκη Φόρντ νομίζω είναι καλοί, καλές προτάσεις στην πλειοψηφία τους. Θέλω να συγχαρώ κι εγώ γιατί είναι εντυπωσιακό το έργο που έγινε. Οι εκατοντάδες τροπολογίες ε, το αποδεικνύουν και το έργο που γίνεται και εξελίσσεται τώρα. Στη δική μου περίπτωση είναι αποδεικτές κάποιες ε, ε, ε, συμβιβαστικές λύσεις. Είναι υποδειγματική η Ισπανία. Η πώληση ε, ε, εκ του μακρόθεν ε, οι τηλεπολίσεις όπλων δεν ευθυγραμμίζονται σε αυτά τα πλαίσια και πρέπει να δούμε ότι σε αυτούς τους συμβιβασμούς πρέπει να δούμε ότι πρέπει να φουγκραζόμαστε συγκεκριμένους τομείς και ομάδες. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ συγχαίρω την κυρία Φόρντ για την εργασία που έκανε γιατί ξεκινήσαμε από ένα κείμενο της Κομισιόν που ήταν απολύτως ε, ε, χωρίς καμία ισορροπία και ε, βεβαίως εμείς θέλουμε ε, να μην να, ασχοληθούμε μονάχα με αυτούς που πραγματικά πρέπει να μας απασχολήσουν όχι δηλαδή τους κυνηγού ή αυτούς που κάνουν αθλητική σκοποβολή γιατί ποτέ οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν ξεκινούν από αυτούς. Τώρα, η αδειοδότηση των πέντε ετών δεν είναι καθόλου χρήσιμη. Θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό γιατί θα, δημιουργήσει, θα δημιουργήσει πρόβλημα στους ε, κυνηγού, αλλά δεν θα ενοχλήσει καθόλου τους ε, ε, τρομοκράτες. Όσον αφορά την πώληση εξ αποστάσεως ή μέσω ίντερνετ πιστεύω ότι οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο φυσικής επαφής. Επίσης θα πρέπει να απαγορευτεί πάντελώς η δυνατότητα αγοράς με ε, Όσον αφορά την σήμανση των κύριων στοιχείων ε, του ε, όπλου. Δεν πρέπει και εδώ να μπερδευόμαστε και να δημιουργούμε εχθρούς χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί υπάρχουν και μερικά στοιχεία που είναι πάρα πολύ μικρά. Τώρα, ξέρετε... Ε, ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε καλά το θέμα της ε, χρονολόγησης γιατί έχουν γίνει τρομοκρατικές επιθέσεις ε, με όπλα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης όσον αφορά την αποθήκευση των όπλων ξέρετε ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αποθηκευτεί ένα όπλο αυτόματο ή με αυτόματο εάν σπάσει στα δύο και αποθηκευτεί το ένα στο ένα σημείο και το άλλο στο άλλο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σάλαχο. Thank you, Chair, and thanks to Mrs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την κυρία Φόρτε για την πολύ σκληρή δουλειά που έκανε. Ε, οι συμβαστικές ε, τροπολογίες είναι πολύ καλές, αλλά θέλω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα. Πράγματι πρέπει να απορρίψουμε την προτινόμενη κατηγορία Α7 αλλά δεν πρέπει να την ξαναφέρουμε ως B7. Ε, δεν χρειάζεται, κανένα κράτος μέλος δεν το εφαρμόζει και αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες απόψεις ε, για την, τον περιορισμό ε, στη διαδικασία της αναγόμωσης, του γεμιστήρα, της, ε, ε, του, της χωρητικότητας του γεμιστήρα και ξέρουμε ότι αυτό έχει δοκιμαστεί ε, σε πολλές ε, χώρες. Η ρυθμοί σχετικά με τον γεμιστήρα, αυτό ε, θα κάνει δύσκολη τη ζωή σε πολλούς. Επίσης θα μεγαλώσει το βάρος στις αρχές που εκδίδουν τις άδειες. Στο άρθρο 10 αναφέρεται και παρατέτω, ο αγορισμός των πυρομαχικών επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν άδεια να αγοράσουν πυροβόλο όπλο από τη σχετική κατηγορία. Νομίζω αυτό βασίζεται σε μία παρεξήγηση. Τα πυρομαχικά δεν προβλέπονται για ένα συγκεκριμένο πυροβόλο όπλο ή κατηγορίες πυροβόλες όπλων. Αυτά είχα να σας πω και σε ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκραπίνη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι η δήμον σε θέματα όπλων. Γι' αυτό και ανησυχώ για τα όσα τεκταίνονται στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια. Είναι πολύ ανησυχητικά τα όσα βλέπουμε να γίνονται γύρω μας. Αληθεύει ότι δεν είναι τα τρομοκρατικά πλήγματα πράξεις κυνηγών για παρεμμένους σκοπευτών, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν δεν έχουμε αυστηρούς κανόνες, τότε θα είναι εύκολη η κατοχή όπλων και μπορούν να σημειωθούν και ατυχήματα. Υπάρχουν τέτοιου είδους πολλά κυνηγητικά ατυχήματα. Θα ήθελα σε τρία σημεία να εστιαστώ. Πρώτον, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση και για τις, ε, ε, τα ιατρικά πιστοποιητικά. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να διοργανωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο για όλους, άσχετα ποια θα είναι η χώρα προέλευσης. Είναι σημαντικό αυτές οι ιατρικές εξετάσεις σε όλα τα κράτη να είναι, θα έλεγα, ταυτόσιμες, να είναι ισότιμες, ώστε να μην μπορεί κάποιος να μετακινείται σε μια χώρα όπου θα υπάρχει ένα πιο χαλαρό τέτοιο καθεστώς εξετάσεων και ρυθμίσεων. Και το θέμα, για παράδειγμα, όσον αφορά και ε, πιο ηλικιωμένους, ε, για παράδειγμα κυνηγού, ε, δεν θα συμφωνούσα με την επέκταση αυτή μέχρι και τα 80. Το θέμα του ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνο για την αποθήκευση όπλων είναι κέρια σημασία. Πρέπει να αποσαφινιστεί ότι θα είναι πάντα ο κάτοχος του όπλου ο υπεύθυνο. παρακαλώ, στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω θερμά την κυρία εισηγήτρια, λέει η κυρία Σαχναλόβα για την πρότασή της και ευελπιστώ, έχω τη βεβαιότητα θα καταλήξουμε σε καλές συμβιβαστικές προτάσεις. Λέω ότι έχει νόημα και είναι σκόπιμο να υπάρχει έλεγχος των κατόχων όπλων και να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το παρεμπόριο την μαύρη αγορά όπλων. Ευχαριστώ για τις καλές ε, συμβιβαστικές προτάσεις ε, με ε, και τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής ως αυθεντική ομάδα συνεργαστήκαμε. Θέλαμε να αντιδράσουμε ώστε να καλυφθούν τα κενά της νομοθεσίας όπου υφίστανται αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό οι πολίτες, τα κράτη-μέλη και οι ανάγκες τους να λαμβάνονται υπόψη. Τρία συγκεκριμένα θέματα θα ήθελα τώρα να αναφέρω. Αφενός έχουμε την κατηγοριοποίηση σε διαφορετικές ομάδες που είναι σημαντικό, για παράδειγμα την κατηγορία Α6 και μετά ρυθμίσεις όσον αφορά τους ε, εμπόρους ε, και όσους ε, συναλλάσσονται με όπλα και οπλισμό. Είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στις πιο ε, αποτελεσματικές ε, ρυθμίσεις και η πληρωμή με ρευστό, με μετρητά είναι σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν σε πολλά κράτη αποδεκτές ε, προτάσεις και αυτές δεν πρέπει να επιβαρυνθούν ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ για μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ η κυρία Τσάρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, κυρία Φόρντ όπως και άλλοι. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το ζήτημα και βεβαίως εδώ κατανοούμε και πόσο περίπλοκο είναι το, η διαδικασία λήψης απόφασης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εμείς λαμβάνουμε υπόψη ε, ιδιαίτερος ε, και ε, νωρίτερα και εγκαιρότερα υπόψη, λέω, τους προβληματισμούς των κρατών μελών. Υπάρχουν ζητήματα όμως εδώ που παραμένουν σημαντικά. Το θέμα των εφέδρων είναι πολύ ουσιαστικό σημαντικός ο ρόλος τους ε, για την άμυνα ορισμένων ε, χωρών. Ε, υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε στην άλλη πλευρά του Αντιλαντικού λένε ότι θα σταματήσουν οι πυροβολισμοί στα σχολεία εάν όλοι οι μαθητές και όλοι έχουν όπλα. αν είναι δυνατόν. Εμείς θέλουμε ευρωπαϊκή απάντηση. Ο κύριος Κάρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν αυτό το πώς εμείς συζητούμε αυτό το ζήτημα εδώ είναι ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα πώς πρέπει ευαίσθητα θέματα να αντιμετωπίζονται απαντούμε στις ευαισθησίες ε, που υφίστανται όχι συναισθηματικά. Αντικειμενοποιούμε τα πράγματα, προσπαθούμε με αντικειμενικό τρόπο να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να καταθέσουμε τροπολογίες. Και αυτό είναι κιόλας ε, κάτι πολύ θετικό της, από πλευράς της εισηγήτριας και των σκιωδών εισηγητών που συνεργάστηκαν και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα και καταδεικνύεται και από την καλή συνεργασία και τη συζήτηση. Παρόλη την καλή προεργασία δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα βέβαια. Αυτό το αναφέρω, το δείχνουν και οι συζητήσεις και οι προτάσεις όσον αφορά και την παρέμβαση Κοφεράτη. Για αυτούς που μας ακούνε πρέπει να πούμε ότι η πρόταση, με την πρότασή μας και τη δράση μας ε, ε, απομακρύνεται, διαγράφεται η πρόταση, ρυθμίζονται τα θέματα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα υπάρξει νομιμοποίηση ε, των, της κατοχής όπλων με κανένα τρόπο ώστε να είναι εύκολη. Επανεπεξεργαζόμαστε την οδηγία για την κατοχή όπλων λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα. Όμως αυτή η οδηγία δεν δίνει απαντήσεις στα τρομοκρατικά πλήγματα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα που έχουμε. Και γι' αυτό χαίρομαι για το ότι υπάρχουν τροπολογίες ε, για την ε, προσθήκη ε, εξετάσεων, για παράδειγμα ιατρικών εξετάσεων που θα προβλέπονται για την κατοχή όπλων. Η κυρία Μέτσολα, ευχαριστώ. Και εγώ προσθέτω τη φωνή μου, ευχαριστώντας την εισηγήτρια και τους χειώδεις εισηγητές για αυτή την προσέγγιση. Και είμαστε υπέρ μιας αυστηρής, ε, ε, ενός αυστηρού ελέγχου κατοχής όπλων ε, για την καταπολέμηση φυσικά και φαινομένων όπως της τρομοκρατίας. Ωστόσο όμως ε, δεν πρέπει να υπάρξει μια ισοπεδωτική αντίδραση. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την συμβαστική τροπολογία 11 που την ε, διασύνδεση νόμιμων κατόχων όπλων και ε, τρομοκρατικών περιστατικών την διαγράφουμε. Για την προσθήκη για τις αναγκαίες ρήτρε ασφάλειας που πρέπει να προβλέπονται και από πλευρά των κρατών μελών τον αναγκαίο ρόλο που πρέπει να αναλαμβάνουν για τα τεχνικά ε, εξαρτήματα και συστατικά ε, ουσιαστικά στοιχεία των όπλων πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις ε, διεθνείς πρακτικές όπως το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών. Μας ανησυχεί το θέμα των πυροβόρων όπλων και πρέπει να δούμε το ποιοι θα κατέχουν τα όπλα. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται οι όπαδοι, οι, όσοι είναι σκοπευτές για παράδειγμα και κυνηγοί και δεν πρέπει με αυτόν τον τρόπο να τους πλήττουμε. Όμπερμαϊερ παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς ε, και με την πρόταση αρχικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε μια λανθασμένη προσέγγιση για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και επιβάρυνε τους ε, σκοπευτές ε, κυνηγού και για παράδειγμα όποιος θέλει να αγοράσει ένα πυροβόλο όπλο θα πρέπει να δει για παράδειγμα ότι σε σχέση με την εξέβρεση όπλων εύκολα σε κάποιες αγορές μπορεί να διασφαλιστεί αυτό. Πρέπει να δούμε σε σχέση με το δίκαιο που υφίσταται σε κάποια κράτη-μέλη τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ε, μπορούμε να υιοθετήσουμε και να ακολουθήσουμε. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι χρήσιμο. Παραδείγματα για αυτά. Η, ε, στην Αυστρία έχουμε σαφείς ε, ρυθμίσεις όσον αφορά τους αδειοδοτημένους πιστοποιημένους εμπόρους όπου υπάρχουν ε, έλεγχοι, μετατροπές ε, μετατροπές σε σχέση με την, ε, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του όπλου πρέπει να είναι αντικείμενο καταχώρησης χωρίς υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση και πρέπει ακριβώς να προσέχουμε να μην εγκληματοποιούμε κάποιες πράξεις χωρίς ε, να υπάρχει λόγος και να μην υπερβαραίνουμε υπερβολικά γραφειοκρατικά τέτοιου είδους ε, διαδικασίες. Και πρέπει να δούμε την ασφαλή αποθήκευση όπλων ε, και οπλικού υλικού που πρέπει να διασφαλίζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και εδώ πάλι χωρίς γραφειοκρατική επιβάρυνση ώστε να εφαρμοστούν αυτά αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπερμάγερ. Σόλτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ε, για εξέβρεση συμβιβασμών η πρόταση της Κομισιόν στην αρχική της ε, μορφή ε, δεν ε, μας ικανοποιεί με την έννοια ότι μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά την καταπολέμηση της, τροπολογ... τρομοκρατίας αλλά δεν κλείνει την ψαλίδα των διαφορετικών προσεγγίσεων από πλευρά των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν εναρμονισμένοι κανόνες που θα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα παντού. Εγώ προέρχομαι από την Σλοβενία όπου ε, η νομοθεσία που αφορά τον έλεγχο των όπλων είναι εξαιρετική και επομένως εμείς δεν θα επιθυμούσαμε να, ε, ε, να την τροποποιήσουμε επιταχύρω. Ε, καμιά φορά, επομένως ε, θα πρέπει όταν ε, προσπαθούμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις θα πρέπει λέω να λαμβάνουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες, να παίρνουμε κάποια καλά παραδείγματα και οπωσδήποτε να μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε συλλέκτες, σε κυνηγούς κτλ. Ο κύριος Βάμπε. Είμαστε σε πίεση χρόνου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους εσκιώδης εισηγητές για όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει. Πράγματι τα 28 κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς κανόνες. Κάπου όλοι αυτοί πρέπει να ε, συνδεθούν και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αναζητήσουμε συμβαστικές προτάσεις. Αλλά ε, ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί δεν θέλουν να γίνει τίποτα στην Ευρώπη, να επιτευχθεί τίποτα. Εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου σε δύο τροπολογίες. Είμαι ευγνώμων ε, για το ότι πολλές από τις δικές μου τροπολογίες συμπεριλήφθηκαν στις συμβιβαστικές, αλλά αναφέρομαι σε δύο. Στην 525 τα κριτήρια για την έκδοση άδειας οπλοφορίας. Και νομίζω ότι η πρόταση που γίνεται είναι πολύ πιο αποτελεσματική από το να μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη ό,τι επιθυμούν. Δηλαδή, αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι ε, δεν καλύπτονται πλέον τα κριτήρια για την ε, άδεια πληροφορία, τότε θα πρέπει να παραμένουν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια ερώτηση και στην Και το δεύτερο ερώτημα αφορά τα ήμια αυτόματα όπλα. Και με ενδιαφέρει γιατί καταλήγουμε στην, ε, στον ορισμό ότι πρόκειται για όπλα που resemble, που μοιάζουν ή προσωμιάζουν με επικίνδυνα όπλα. Γιατί αυτό. Ε, πρόκειται για είναι αυτόματα όπλα, τα οποία όμως μπορούν να μετατραπούν σε πλήρως αυτόματα όπλα. Αυτά θα ήθελα να ρωτήσω και νομίζω ότι κατά τα άλλα μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Έχουμε εδώ κοντά μας εκπροσώπηση του Συμβουλίου. Πριν λοιπόν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για την τελική της παρέμβαση, θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στους εκπροσώπους ε, της Επιτροπής, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι, κατά το μέγιστο δύο λεπτά χρόνος ομιλίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι και εσείς κάνατε τις ίδιες συζητήσεις που κάναμε και εμείς. Την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, η Ολλανδική Προεδρία ε, πέτυχε μία ισορροπημένη προσέγγιση σχετικά με την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Εμείς είμαστε πολύ πιο αυστηροί για τα πυροβόλα όπλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γρήγορα θα σας πω και κάποια παραδείγματα. Ε, νέοι κανόνες ε, σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους, ε, το πώς θα εντοπίζονται για να μπορεί να βελτιώνεται η ίχνη λασιμότητα. Επίσης, για να υπάρχει σαφής ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη ορίσαμε τους συλλέκτες και αυτοί καλύπτονται από την επιγεία, αυτοί καλύπτονται από αυστηρές συνθήκες ασφαλείας. Ε, πρέπει να απαγορεύονται τα επικίνδυνα ε, ημιαυτόματα όπλα και να υπάρχει αυστηρότερο ε, καθεστώς για ακουστικά όπλα και για όπλα χαιρετισμού salute weapons and acoustic weapons. Είναι σημαντικό λοιπόν σύντομα να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος και να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο για την τελική εισήγηση στην κυρία Φόρντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάποια θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και από άλλους. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στο θέμα των ε, συλλεκτών και των μουσείων. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί σε κάποιους οργανισμούς ότι κοίταξε εσύ είσαι μουσείο και εσύ δεν είσαι, είσαι συλλέκτης. Γιατί σαφώς και υπάρχουν κάποιοι φορείς που είναι στη μέση αυτών των δύο. Και είναι σημαντικό το ότι και αυτοί που είναι ιδιώτες ε, συλλέκτες και για αυτούς ε, να υπάρχουν σαφείς κανονισμοί, ασφαλής αποθήκευση και να έχουν συλλογές μόνο αν πραγματικά συλλέγουν για ιστορικούς ε, σκοπούς και μόνο εφόσον η συλλογή διατηρείται σε ένα επίπεδο που δεν θέτει σε κίνδυνο την δημόσια ασφάλεια. Όλα αυτά βρίσκονται στη συμβαστική πρόταση. Όλα αυτά βρίσκονται στη συμβαστική πρόταση. Όσον αφορά το θέμα των ιατρικών ε, τεστ, τεστ υγείας. Εγώ έχω πολλούς ε, με ειδικέ ανάγκες ε, που μου υπενθύμησαν ότι είναι παραολυμπιακοί ε, βολής που... Ε, α, που Επίση, κάποιοι με ειδικέ ανάγκε που δεν ακούν καλά χρησιμοποιούν όπλα ακουστικά που δεν βλέπουν, ναι, ναι που δεν βλέπουν καλά, τα χρησιμοποιούν για να ακούνε την ε, τροχιά που ακολουθεί το βλήμα. Όλοι λοιπόν πρέπει να έχουν ένα σύστημα διότι κανείς ε, δεν που αποτελεί κίνδυνο για το κοινό και τους συμπολίτες του ε, δεν μπορεί να έχει άδεια πλοφορίας. Όποιος είναι επικίνδυνος δεν μπορεί να παίρνει αδειο Και αυτό δεν οφείλεται ή δεν κρίνεται από το κατά πόσο είναι κανείς αρτιμελής ή όχι. Καμία σχέση. Κάθε χώρα πρέπει να έχει τις δικές της διαδικασίες, να είναι σαφείς και άκαμπτες και πρέπει να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα. Όσον αφορά τα πυρομαχικά, οι τροπολογίες μου έχουν ως στόχο ότι να απαγορεύσουν να σωρεύει κανείς ε, πυρομαχικά. Ας πούμε, αν έχει κανείς ένα όπλο, γιατί αγοράζει πυρομαχικά για τελείως διαφορετικό τύπο όπλου. Τώρα, για τα ημιαυτόματα όπλα. Το κείμενο του Συμβουλίου έρει τα ημιοαυτόματα που έχουν μετατραπεί από αυτόματα. Όμως επαναφέρει την άδεια σε κάποιες περιπτώσεις στη σκοποβολή. Και λένε κάποιοι ότι αυτό αν είναι σε επίπεδο μόνο κράτους μέλους, δεν μπορούν όσοι ασχολούνται με αυτό το άθλημα να πάνε να συμμετέχουν σε αγώνες σε άλλη χώρα. Άρα δηλαδή ελπίζω να ψηφίσουμε για κάθε ένα από αυτά τα διαφορετικά θέματα να επιτύχουμε κάποια πλειοψηφία και μέσα από τον τριμερή ε, διάλογο να επιτύχουμε μια σαφή διατύπωση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Πριν ολοκληρώσουμε την ε, ευρύτατη αυτή συζήτηση, ότι η δεύτερη συζήτηση για τις συμβαστικές τροπολογίες θα λάβει χώρα την 13η Ιουλίου και ότι στις 14 Ιουλίου, σημαντική ημερομηνία, θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ σας ευχαριστώ πολύ. Um, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα έχουμε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων Θα έχουμε λέω ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο κυρία Βέρα Γιουρόβα Ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρία Επίτροπε, και ε, με ρώτησαν «Μα γιατί φεύγεις τώρα και πας στις Βρυξέλλες» και είπα «Μα γιατί θα έρθει η, εκπρόσωπο, η Επίτροπος ενώπιον του Κοινοβουλίου για να μας πει περί τίνος πρόκειται και τι έχει κάνει». Και μου είπαν «Α, μα δεν είχαμε καταλάβει ότι το Κοινοβούλιο έχει τέτοια εξουσία». Μα αυτό είναι ακριβώς ε, η δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπόλογος ενώπιον του Κοινοβουλίου στα πλαίσια αυτής της ε, δημοκρατικής διαδικασίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που είσαστε εδώ μαζί μας να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα της Κομισιόν. Η Επίτροπος θα μιλήσει για περίπου 20 λεπτά και μετά θα δεχθεί ερωτήσεις. Έχουμε πολλές ε, ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο βέβαια πρώτα στους συντονιστές και μετά στους υπολείπους. Ε, θέματα καταναλωτών λοιπόν θα μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ α, για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κανάλτες. Έχουμε αρκετά θέματα υπό προπαρασκευή ώστε να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο για το μέλλον. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω μια επισκόπηση των προτάσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα και τα μελλοντικά μας σχέδια το δίκαιο για την προστασία καταναλωτών ε, έχει εξελιχθεί ταχύτατα κατά τα τελευταία χρόνια με την οδηγία για τα δικαιώματα καταναλωτών, ε, για τα θέματα τα ψηφιακά και για την προστασία και τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών, αντιμετώπιση των αθέμητων πρακτικών μέσα από την σχετική οδηγία, όλα αυτά έχουν κοινό στόχο να καλυφθούν τα κενά και να αναγνωρίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών. Και όσον αφορά το μέχρι σήμερα κεκτημένο, το οποίο υφίστατο επί σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφάσισα να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε σε έξι ε, συνιστώσεις τα όσα έγιναν ε, για την ε, πρακτική τους εφαρμογή και αποτελεσματικότητα. Να είναι απόλυτα σαφές. Στόχος δεν είναι να καταργηθούν κείμενα για την προστασία των καταναλωτών, αλλά η μείωση γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε τη δουλειά αξιολογώντας τι λειτουργεί καλά, τι πρέπει να εξυγχρονιστεί για το μέλλον και πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει πιστοποίηση κανονισμών, εκεί όπου δεν χρειάζονται θα ε, εξαλείφθουν, θα διαγράφονται, πέρα από αυτή την αναδρομική αξιολόγηση και εξέταση για τους καταναλωτές, θέλουμε να έχουμε και τις απόψεις των εμπλεκομένων με τις απόψεις τους ε, για την ε, βελτιστοποίηση και τον εξυγχρονισμό. Ιδιαίτερα θέλουμε πρώτον θέματα καταναλωτών στην ε, πολυμερή οικονομία να λαμβάνονται υπόψη να λαμβάνουμε υπόψη τα θέματα, για παράδειγμα, όπως του περιβάλλοντος, να βελτιώσουμε την ε, επικοινωνία και τις πληροφορίες που θα διαχέονται προς τους καταναλωτές και τελευταίο που θέλω να το τονίσω αυτή τη στιγμή είναι ένα πιο ενδυναμωμένο, ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, <clears throat> αντιμετώπιση οποιασδήποτε ε, ζημίας ή βλάβης βάρος των καταναλωτών. Από τον Μάιο στο Σεπτέμβριο είναι η διάρκεια αυτού του εγχειρήματό μας και πραγματικά σας ζητώ να ε, προσπαθήσετε να διαδώσετε στο μέτρο του εφικτού αυτά τα στοιχεία. Έχουμε επίσης ε, και μια ομάδα των εμπλεκομένων ενδιαφερομένων με ΜΚΟ που θα μπορέσουν να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Αυτό ο έλεγχος θα είναι το κοινό στοιχείο για την Σύνοδο Κορυφής για θέματα καταναλωτών κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ένα ευρύτατο φάσμα εκπροσώπων και πραγματογνωμόνων που θα προσέλθουν στις Βρυξέλλες για να εξεταστεί η μελλοντική αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων υπέρ των καταναλωτών. Θα ε, την ενεργό συμμετοχή σας σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα ψηφιακά έχουμε επιταχύνει την ανάλυση όσον αφορά την εξέταση ε, σε σχέση με πωλήσει ε, και την οδηγία σχετικά. Αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο και θα σας γνωστοποιηθούν από πλευράς μας ε, τότε. Ίσως θα έπρεπε επίσης να αντιμετωπιστούν και τα, όσα σας ενδιαφέρουν, τα μελήματά σας, να φύστανται κοινοί κανόνες και ρυθμίσεις για καταναλωτές για τα δικαιώματά τους για παράδειγμα όπως ε, προαναφέρθηκε για τις ε, κοινέ αυτές ε, προδιαγραφές από τα αποτελέσματα και συμπεράσματα αυτού του κοινού έργου και αξιολόγησης θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε την ευθυγράμμιση των κανόνων και κανονισμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο <clears throat> και να διασφαλιστεί και η πρόσθετη αξία που ε, θα μπορεί να απορρεύσει. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένων των, ε, δεδομένης της πραγματικότητας της αγοράς σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί στις ηλεκτρονικές πωλήσει και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το ότι ξεκίνησε το έργο του παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αφενός για το ψηφιακό περιεχόμενο και τις ε, ρυθμίσεις αφετέρου. Είναι μια κοινή δέσμη μέτρων και διαδραματίζουν και τα δύο στοιχεία στοιχεία, τον ρόλο τους ε, για τα θετικά αποτελέσματα της ε, ευρωπαϊκής εσωτερικής ψηφιακής αγοράς. Ε, είμαι ευγνώμονα για την θετική ανταπόκριση από πλευράς των αντιδράσεων, από πλευράς εισηγητών και στην Νομική Επιτροπή και στην δική σας Επιτροπή. Βρισκόμουν σε έναν όροφο πάνω από αυτόν στον οποίο είμαστε σήμερα και είχα συζητήσει σχετικά με, τις, ε, ε, ε, το, να ακούσω τις απόψεις των εμπλεκομένων. Αυτοί, αυτές οι προτάσεις πρέπει να διασφαλίζουν μια ισορροπία. Χρειάζονται για την προστασία των καταναλωτών και για την αγορά αυτές οι βέλτιστες προδιαγραφές. Με ένα στοχοθετημένο, προσιλωμένο τρόπο για μια, έναν εναρμονισμό που θα πρέπει να διασφαλιστεί όπως επιθυμούμε δίνουμε συνέχεια στο να υπάρξει ένα ε, σε ανώτατο επίπεδο ε, ε, πλαίσιο ε, για την ε, διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών, πρέπει να λάβουμε από την άλλη πλευρά και την ε, συνιστόσα του εμπορίου και να δούμε ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πωλήσουν περισσότερο διασυνοριακά αν αυτό θα απαιτεί το να γινόταν στο υψηλότατο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο και αν θα μπορούσε να υπάρξει μια σύγκληση επ' αυτών. Οι προτάσεις ε, που έχετε μπροστά σας ε, στοχεύουν στο να υπάρξει αύξηση του πλαισίου ε, προστασίας των καταναλωτών στο δυνατόν υψηλότερο επίπεδο και αυτό εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο την ιδέα της λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς. Πιο εξειδικευμένα στρέφομαι σε αυτές τις προτάσεις τώρα. Στις 25 Μαΐου, όπως γνωρίζετε, υιοθέτησε το πακέτο μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και την αναθεωρημένη ρύθμιση για την προστασία των καταναλωτών κύριο στοιχείο για την ε, υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ακόμα όμως και οι καλύτερες προτάσεις παραμένουν ε, κενός λόγος αν δεν εφαρμοστούν σωστά. Ε, γι' αυτό η πρότασή μας είναι ένας μηχανισμός να αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις και παραβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ενδυναμώνονται, ενισχύονται οι εξουσίες και αρμοδιότητες ώστε να καταπολεμήσουμε διασυνοριακά τις αθέμητες καλές πρακτικές ε, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσει στο ηλεκτρονικό, στο διαδίκτυο εμπόριο για να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε και να αναχαιτήσουμε το δυνατόν ταχύτερα τέτοιου είδους παραβάσεις και παραβιάσεις. Και σε σχέση με ενώσεις και συλλόγους ε, εμπόρων θα διαδραματίσουν και τον ρόλο τους όσον αφορά την ε, αρρωγή σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων συνιστώ να υπάρξει επιλογή αρμόδιου εισηγητή από πλευρά τη Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής ώστε να υπάρξει συμμετοχή στην συνομοθετική διαδικασία. Έχουμε και την πτυχή της πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αθέμητων πρακτικών. Και σε σχέση με την δέσμη μέτρων της 25ης Μαΐου υπάρχει και η αναθεωρημένη επικαιροποιημένη μορφή για την οδηγία αυτών των φαινομένων. Εντοπίζει μετά από ενεργό ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, των τάσεων σε σχέση με το εμπόριο και των επιχειρήσεων ε, ηλεκτρονικά και τις πλατφόρμες κοινωνικού περιεχομένου. Επίσης εξειδικευμένα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εμπόριο σε σχέση με χρήσεις, με χρήστες ακροατές ίσως ε, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα ε, πολύ εμπορευόμενοι. Και αυτό σε σχέση και για την ε, οδηγία κατά του του εμπορίου θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη στη συνάφειά τους. Να προσθέσω μερικά σχόλια για την επιμερισμένη οικονομία υπενθυμίσαμε στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία από τις αθέμητες πρακτικές μέσα σε αυτήν την ενρευστό διαδικασία όπου όλα μεταβάλλονται ταχύτατα είναι ιδιαίτερη προτεραιότητα στο έργο μας και με ανησυχία διαπιστώνουμε ότι υπάρχει βραδύτατη πρόοδο σε σχέση με το Συμβούλιο. Ε, ε, ευελπιστούμε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις επαφές σας και την επιρροή σας σε σχέση με τα κράτη-μέλη ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά και την ασφάλεια. Θα βελτιώσουμε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα. Στρεφόμαστε προς τους εμπλεκόμενους της αγοράς ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, του εμπορίου online. Υπήρξε θετική ανταπόκριση από πλευρά σου. Στο 2015, 62% ε, των επικίνδυνων ε, προϊόντων μέσω του Rapid Eye συστήματος προερχόντουσαν από την Κίνα θα μεταβώ στην Κίνα ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η συνεργασία μας με τις κινέζικες αρχές στον τομέα της ασφάλειας. Μέρος της επίσκεψής μου θα αφορά την, ε, ε, τη Σύνοδο Κορυφής ε, για την προστασία των καταναλωτών με τους εταίρους μας των ΗΠΑ και της Κίνας και τη συμμετοχή φυσικά της ΕΕ ώστε τα θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών να μπορέσουν να καλυφθούν επαρκώς. Κύριε Ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, ευελπιστώ ότι θα εξελιχθεί θετικά η συζήτηση και η επαφή μας και όλα τα θέματα καταναλωτών θα μπορέσουν να καλυφθούν όπως πρέπει. Ευχαριστώ each of the... um... Πολύ ωραία. Ε, θα ακούσουμε λοιπόν τους συντονιστές και τους αντιπροέδρους και μετά ε, θα λάβουμε ερωτήσεις ε, από τα άλλα μέλη. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις ε, νομοθετικές αποφάσεις που έχετε λάβει και αυτά που προτίθεστε να αποφασίσετε. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή η δική μας θεωρεί το refit είναι μεγάλη προτεραιότητα γιατί εμείς πιστεύουμε ότι Όσον αφορά το θέμα το ψηφιακό ή αναλογικό, θέλουμε αυτό να το αποφύγουμε και το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητα του ψηφιακού ή του αναλογικού. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως την πρόταση για το refit και χαιρόμαστε που μας είπατε ότι θα υπάρξει σύντομα η πρόταση αυτή. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο, πιστεύω ότι η πρόταση του ευρωπαϊκού πτωχευτικού δικαίου είναι πολύ σημαντική και για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Διότι αυτό το πτωχευτικό δίκαιο είναι πολύ σημαντικό για πολλά και η λειτουργία της ενιαίας αγοράς αφορά και σε θέματα που έχουν σχέση ε, με τα εχέγγυα με την ασφάλεια ή ανασφάλεια σε διασυνοριακές αγορές. Σε ορισμένους λοιπόν τομείς έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση διότι δεν δανειοδοτούνται από τις τράπεζες επειδή οι τράπεζες δεν γνωρίζουν κατά πόσο είναι εξασφαλισμένα τα υποχωρήγηση δάνεια. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό οδηγεί σε μειονεκτική θέση των ε, κάποιων κρατών μελών. Το πτωχευτικό δίκαιο είναι πολύ σημαντικό και διερωτώ με κατά πόσον έχετε να πείτε κάτι από αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Και πρέπει να σας πω όμως ότι, ξέρετε, μπερδεύτηκα λιγάκι. Καλό το refit. Πολύ καλό το fitness check. Και ε, στόχος είναι βεβαίως ε, να υπάρχει συνέπεια στην ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να υπάρχουν απλουστεύσεις όπου είναι αυτό δυνατό και να διατηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Όλα αυτά καλά και ωραία. Όμως δεν κατανοώ της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί με αυτές τις πράξεις φτάνουμε στο ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικές προτάσεις για το offline και το online σχετικά με τα καταναλωτικά αγαθά που σημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος ανάλογα με το κατά πόσο να έχει αγοράσει κανείς ε, ένα αγαθό διαδικτυακά ή όχι από εκεί οι εταιρείε στο τέλος να μην γνωρίζουν καν ε, σε ποια ακριβώς ε, διαδικασία βρίσκονται. Άρα δηλαδή εδώ ολοχεύει ένας κίνδυνος, ουσιαστικός κίνδυνος ασυνέπειας και ε, εσείς ε, απευθύνεστε στο Κοινοβούλιο ε, και θέλετε όλα αυτά να αντιμετωπιστούν ως πακέτο. Εμείς συμφωνούμε, αλλά ξέρετε, να σας πω ότι δεν κατανοώ πια τον τρόπο αντιμετώπισή σας. Κυρίως μετά από αυτά που μας είπατε σήμερα. Μία άλλη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ε, βλέποντας τις ε, προτάσεις, κυρίως όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο, ξέρετε, για την προστασία του καταναλωτή πρέπει να υπάρχει και ουσιαστική προστασία των δεδομένων. Εξ όσων όμως γνωρίζουμε υπάρχουν τεράστια κενά, ε, κυρίως στο άρθρο 3.1. Εκεί γίνεται λόγος για περαιτέρω δεδομένα. Μα ποια είναι αυτά τα περαιτέρω, τι είναι περαιτέρω δεδομένα. Ξέρετε, τόσο ε, ασαφές νομοθετικό κείμενο ε, δύσκολα να δει κανεί. Έχουμε πάρα πολλά για να συζητήσουμε και να διαβουλευτούμε και επ' αυτού και η τελευταία μου ερώτηση. Το refit, καλό. Καλό, μια χαρά το refit. Αλλά σας ερωτώ, οι προτάσεις σας για το δεύτερο εξάμεινο του 2016, ποιες ακριβώς είναι, αυτό θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ, για να γνωρίζουμε, έστω και κατά προσέγγιση, τι έχουμε να περιμένουμε ε, κατά τους επόμενους μήνες της κοινοβουλευτικής μας εργασίας. Dan Dalton. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να φύγω δυστυχώς ε, γιατί ε, έχω να μιλήσω σε, κάποιο, σε μια ομάδα αναποφάσεις των Βρετανών ψηφοφόρων που επισκέπτονται εδώ. Εν πάση περιπτώσει όσον αφορά ε, την μεριστική οικονομία, τη συνεταιριστική οικονομία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και ε, συμφωνούμε ότι ε, αυτού του είδους, με τη δήλωση που λέει ότι αυτού του είδους η συνεταιριστική οικονομία θα είναι η τελευταία προσφυγή και θα πρέπει να διαγραφεί τελευταία, αλλά βλέπουμε αποφάσεις στη Γαλλία και στη Γερμανία σχετικά με την Uber που, Uber που πηγαίνουν προς την άλλη κατεύθυνση. Επομένως αυτή η ίστατη προσφυγή δεν ισχύει. Είχαμε πει ότι με αυτόν τον τρόπο, σαν ίστατη προσφυγή θα μπορούσε να ασχοληθεί να διαγράψει αυτές τις εταιρείε ε, το κράτος. Ε, εμείς ε, πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους διαδικασίες δίνουν δύναμη στο, στους καταναλωτές και πρέπει να τις στηρίξουμε. Οι προτάσεις όμως οι οποίες αναφέρεται θα, δώσουν, θα προκαλέσουν μεγάλο βάρος σε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε άλλες μικρές επιχειρήσεις και επομένως ερωτώ με αυτού του είδους τις συμβάσεις ποιο πρόβλημα προσπαθείτε να λύσετε το πρόβλημα της μη ασφάλειας ας πούμε των στοιχείων γιατί φοβούνται οι άνθρωποι να δώσουν τα στοιχεία τους στο ίντερνετ ε, και κάτι άλλο ε, όσον αφορά την αλληλουχία ε, γιατί πριν από το Refit έχουμε αυτού του είδους τις προτάσεις και πριν λύσουμε τα προβλήματα της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε μια καλύτερη νομοθέτηση νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την ισχύουσα και να εφαρμόσουμε σωστά την ενισχύουσα πριν πάμε σε νέα νομοθεσία. Ευχαριστώ ε, πολύ, λέει η κυρία Σαρανζόβα, ε, κυρία Επίτροπε που ήρθατε εδώ και μας παρουσιάζετε την εργασία σας. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί βλέπω ότι δουλεύετε πολύ για το ψηφιακό θεματολόγιο έτσι ώστε να δώσετε συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί έχουμε αργήσει πολύ. Πρώτον, όσον αφορά το REFIT, ε, να ε, ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τους προηγούμενους ομιλητές. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η μελέτη των ψηφιακών φακέλων. Δεύτερον, ο ε, κανονισμός ε, για την προστασία των καταναλωτών που αναφέρατε. Μπορείτε να μου πείτε πρακτικά πώς βλέπετε το θέμα, γιατί βεβαίως γνωρίζουμε ότι αν υπάρχει καλύτερα και μεγαλύτερη συντονισμένη δράση είναι κάτι αποφελές ε, ε, ε, έχει σαν αποτέλεσμα και εξοικονόμηση πόρων, αλλά πρακτικά πώς μπορείτε να το δείτε αυτό, υπάρχουν οι μηχανισμοί ήδη, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν δεν θα είναι ιδιαίτερος βαριές τελευταία, αλλά πολύ σημαντική παρατήρηση επίσης όσον αφορά τις πλατφόρμες η ανακοίνωση για τις πλατφόρμες ήταν ενδιαφέρουσα ε, και ε, διάβασα ανάμεσα στις γραμμές ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα τροποποιηθεί. Ωστόσο τώρα ε, ακούω φήμες ότι θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά τις, τη συμβατική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές. Μήπως μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι δεν ισχύουν ή ότι ισχύουν ενδεχομένως οι σε αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι θέλουμε να αποφύγουμε παρεκκλήσεις όσον αφορά τους κανόνες και κανονισμούς για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για το κανονικό εμπόριο. Και ταχύτητα χρειάζεται επίσης ώστε να μπορέσουμε σε σχέση με τις ψηφιακές προτάσεις να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για τους καταναλωτές. Αλλά για να είμαστε συνεκτικοί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα σε ένα κοινό πλαίσιο. Θα ήθελα να γνωρίζω αν στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για το πώς το ψηφιακό περιεχόμενο θα μπορέσει να βαίνει εκ παραλίλου με, τις, ε, με το περιεχόμενο της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων και το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Ε, δεν είναι τόσο απλό να αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα ως ένα τρέχον θέμα. Πολλά θέματα εμπλέκονται εδώ. Δεν είναι λοιπόν αυτό ε, θέμα ιδιοκτησίας και η προστασία των δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε ε, οι καταναλωτές να μην καταλήγουν σε μια κατάσταση αθέμητου ανταγωνισμού όπου θα βρίσκονται σε αρνητική θέση όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία θα πρέπει να γνωστοποιούνται όσον αφορά ένα πλαίσιο συναλλαγής. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στην πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο ε, θα πρέπει όπως και στην άλλη πρόταση να έχουμε ένα πλαίσιο αντικειμενικής προστασίας των καταναλωτών και η συμβατική σχέση αυτή να μπορεί να διαμορφωθεί σε σχέση με τους καταναλωτές και τους παρόχους στο πιο ενδεδειγμένο πλαίσιο. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης και στο θέμα της μονοπρόσωπης εταιρεία. θέμα το οποίο εξετάσαμε στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή πριν από τις, ε, τη γνωστοποίηση των εγγράφων Παναμά και των στοιχείων από τον Παναμά και σε σχέση με την ρύθμιση ώστε να μην υπονομεύεται η διαφάνεια, να μην γίνεται όχημα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής η μονοπρόσωπη εταιρεία. Και πραγματικά λοιπόν ε, πώς στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό να το αποτροχοπεδίσει ώστε να ευδοκιμήσει. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Καμιά από τις άλλες ομάδες ε, ζήτησε, δεν παρίσταται για να παρέμβει θα έχουμε και παρατηρήσεις και ερωτήσεις από πλευράς αντιπροέδρων. Εγώ κανονικά θα ρωτούσα την τελευταία, θα ήθελα την τελευταία ερώτηση, όμως σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια εξαίρεση. Επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς χρησιμοποιούν αλγορίθμους ώστε τέτοιου είδους ε, προϊόντα σε σχέση με τους καταναλωτές να μπορέσουν ε, να προαχθούν και χρησιμοποιούν και big data, δηλαδή μεγαστοιχεία. Θα πρέπει να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπίζονται από πλευράς καταναλωτών ομαδοποιημένα σε σχέση με τις ε, προσφορές. Υπάρχουν όμως πολλές ηθικές επιπτώσεις ε, και σοβαρές επιπτώσεις. τέθηκε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν σε σχέση με το Google να γνωρίζει κάποια στοιχεία προτού έχει γνωστοποιηθεί αυτό στους γονείς μου. Και ένα πρόσφατο παράδειγμα, μία ας το πω έτσι τρομοκρατικής ε, προσέγγισης ε, ε, εξέτασης σε σχέση με πρόσφυγες που βρισκόντουσαν στην Ελλάδα με τεχνική ανάλυση αλγορίθμων και προσωπικών στοιχείων. Πώς θα δημιουργήσετε τέτοιου είδους ε, περιβάλλον ώστε με τους αλγορίθμους ε, ο περίγυρος ε, και οι διατάξεις να είναι συμβατές και να συνάδουν με τις προδιαγραφές και τις ρυθμιστικές διατάξεις και νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Η Μαρία, ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει κυρία Κοράτσα την ε, προθυμία και διαθεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με ανησυχεί το θέμα των παιδιών ως καταναλωτών και νομίζω αποτύχαμε να προστατεύουμε τα παιδιά ε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αλλάξει απλώς το επίπεδο ηλικίας όσον αφορά τα φίλτρα και την ε, ε, προστασία από πλευράς ε, των ρυθμίσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το ότι έχετε συνειδητοποιήσει την τεράστια πρόκληση αυτή για τα παιδιά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο διαδίκτυο στο διαδίκτυο και είναι μια προτεραιότητα για μένα αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ο διαχωρισμός μεταξύ της ε, προσέγγισης ε, προστασίας καταναλωτών ηλεκτρονικά και εκτός ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλα όσα προσπαθήσαμε να κάνουμε πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια αμερόληπτη τοποθέτηση. Είναι ένα εργαλείο το διαδίκτυο και εδώ επηρεάζεται η σχέση αγοραστή και πολιτή ε, στη συναλλαγή αυτή και πρέπει να στοχεύουμε στο να προστατέψουμε τους καταναλωτές. Στόχος μας πρέπει να είναι ο πλήρης εναρμονισμός της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και ηλεκτρονικά και εκτός ηλεκτρονικού ε, πλαισίου. Τι θα γίνει με το refit λοιπόν για τα ηλεκτρονικά δικαιώματα, για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε αυτό το πλαίσιο, το εναρμονισμένο πλαίσιο. Υπάρχει εδώ επικέντρωση περισσότερο στην υποχρέωση να ε, προάγονται οι πωλήσει ε, και πρέπει να δούμε εδώ σε σχέση με τη διαφοροποίηση αυτό το θέμα. Πρέπει εδώ όμως να ευαισθητοποιήσω το ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι τόσο η λύση την οποία έχω έτοιμη για να προτείνω και η τελευταία ε, παραγωγή παρατήρηση αφορά την επιμεριστική οικονομία, collaborative economy και πρέπει να δούμε τι θα μπορεί να γίνει με τις πλατφόρμες. Σε σχέση με την καινοτόμο προσέγγιση στην ψηφιακή επανάσταση ελπίζω ότι δεν θα υπερβαρύνουμε υπερβολικά με τις ρυθμίσεις μας αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Euh, Επόμενος αγορητής, σας ευχαριστώ. Επίτροπε, σας ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για τα σχόλια. Νομίζω συμφωνώ και ένα θέμα, μια ερώτηση που θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα που κάνατε, ε, αναφέρατε στο τέλος της δήλωσής σας, ε, όταν αναφερθήκατε στα επικίνδυνα προϊόντα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε, προέρχονται από την Κίνα. Θα πάτε, είπατε, στην επόμενη εβδομάδα στην Κίνα. Υπάρχουν όμως ε, και προηγούμενα σε σχέση, για παράδειγμα, με τον συναγερμό του 2015, 2.000 προϊόντων που δεν ήταν μόνο παιδικά παιχνίδια, αλλά ε, πάσης φύσεως αντικείμενα σε κάποιο σημείο μιλήσατε και είπατε ότι υπάρχει απουσία προόδου και πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ε, να αναζητηθεί διέξοδος από αυτό το αδιέξοδο. Σε σχέση με τους ευρωβουλευτές ε, ζητήσατε να ασκήσουν την επιρροή τους στα κράτη-μέλη ώστε να αποτροχοπεδηθούν τα πράγματα. Εδώ νομίζω όμως ότι το αντίθετο θα πρέπει να υιοθετήσουμε ως προσέγγιση. Για το Google για παράδειγμα αναφέρθηκε προηγούμενα η περίπτωση Google. Όταν ένα κράτος μέλος αρχίζει να ε, ε, ασκεί μια πιο επιθετική πολιτική σε σχέση με τις, ε, τα θέματα αυτά. Και όταν βρισκόμαστε στο θέμα της Κίνας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που παρισφρέουν στην αγορά, αν θα μπορούσαμε σε σχέση με 500 εκατομμύρια καταναλωτές να δούμε αυτή την συνιστόσα και τα παιχνίδια τα οποία εισάγονται από την Κίνα δεν θα ήταν δεν θα είναι δυνατόν να παραμείνουμε αδρανείς. Όταν έχουμε το θέμα των επικίνδυνων προϊόντων, δεν είναι μόνο ένα εξειδικευμένο πεδίο εξειδικευμένων προϊόντων. Έχουμε και το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο να υφίστανται όλο και περισσότερες πωλήσει, να διεξάγονται όλο και περισσότερε πωλήσει ε, με τέτοιου είδου ε, επικίνδυνα προϊόντα. Και με την οικονομία Σέγγεν ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, ε, μπορούν τέτοια προϊόντα να ε, καταστούν επικίνδυνα. Και όταν έχουμε το θέμα της αύξησης ε, της ε, ηλικίας της υπεργύρανσης ε, του πληθυσμού και έχουμε αύξηση αριθμού ατόμων που έχουν ειδικέ ανάγκες πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα αυτά θα είναι ασφαλή και δεν θα υπάρξει βλάβη η ζημιά που θα προξενείται σε κάποιον που θα είναι πιο ηλικιωμένος. Μια λοιπόν αυτή ε, απλή ερώτηση πριν φύγετε και πάτε στην Κίνα. Τι θα ζητήσετε από τους Κινέζους. Θα τους πείτε η Ευρώπη δεν θέλει, δεν επιθυμεί τέτοιου είδους προϊόντα να εξάγονται σε αυτήν. Τι είδους λοιπόν βήματα και διαβήματα θα κάνετε και τι θα απαιτήσετε από τους Κινέζους ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. would you like to ask Ο Νίκολα, <clears throat> κοιτάξτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όλο αυτό το πακέτο της νέας αγοράς της ψηφιακής, όλο αυτό θα λειτουργήσει εάν προστατεύουμε τους καταναλωτές. Ε, μπορούμε να δούμε τα στοιχεία και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα η απαραίτητη εμπιστοσύνη για να, γίνει, ε, για να γίνουν επενδύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Λίγες εταιρείε πουλάνε ηλεκτρονικά και κατόπιν οι καταναλωτές αγοράζουν ε, προϊόντα όπου ο κίνδυνος είναι αρκετά περιορισμένος. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι από τη δυνατότητα να προσφέρουμε προστασία να προστατεύουμε τους κατανοητές, από εκεί εξαρτάται και το κατά πόσον θα μας δοθεί η δυνατότητα να προστατεύσουμε πλήρως την ενιαία ψηφιακή αγορά. Εγώ λοιπόν ε, εύχομαι η πρόταση που έγινε από την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, αυτό να αποτελέσει αφορμή για να φτάσουμε σε μια πιο αυστηρή κατάσταση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και με τον τρόπο αυτό ε, να τηρήσουμε όλες τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπετε για το ψηφιακό εμπόριο. Και τέλος πιστεύω ότι υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο ε, το οποίο ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να έχουμε ουδέτερη επιτροπή. Το θέμα του κανονισμού για τον έλεγχο και κυρίως για το made in. Ε, το Κοινοβούλιο εξέφρασε σε ψηφοφορία την προηγούμενη εβδομάδα την άποψή του και νομίζω ότι η Επιτροπή πριν αρχίσει να σκέπτεται κανόνες οι οποίοι θα αποκλείσουν ε, συγκεκριμένες ε, προβλέψεις όπως το άρθρο 7, η Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί έτσι ώστε να καταλήξει σε σοβαρό και ουσιαστικό συμβιβασμό ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ε, θα έλεγα η Επιτροπή να απαντήσει τώρα και μετά θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Δέκα λεπτάκια five more, or do you want? leave after 12. <laughs> Thank you. So what Ωραία. Ε, να απαντήσετε λοιπόν σε ερωτήσεις που ακούσατε μέχρι τώρα και μετά να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που με υποβάλλατε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και για τις παρατηρήσεις ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δούμε ποιο είναι το κυριότερο ζήτημα το οποίο αναφέρεται στο online και offline στις συναλλαγές. Κατανοώ απόλυτα κυρία Εύελιν Γκέπχαρτ ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σύγχυση σε εσά και σε άλλους και δεν είναι αυτό το οποίο εμείς στοχεύσαμε. Δηλαδή κάποιος που τόσο σε βάθος εμπλέκεται και είναι εξοικειωμένος με θέματα προστασίας καταναλωτών πρέπει να μπορεί να βοηθηθεί. Θέλω να δραχθώ τις ευκαιρίες και να επεξηγήσω πώς εννοούμε τα πράγματα με αυτές τις δράσεις μας. Να δημιουργηθεί ή να καλυφθεί μόνο η πτυχή των ηλεκτρονικών συναλλαγών υπό την οδηγία ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και σας το είπα και την τελευταία φορά ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε το θέμα της στοχοθετημένης, του στοχοθετημένου εναρμονισμού για κανονισμούς και διατάξεις όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για τις ε, κατά το παρελθόν προσπάθειες που είχαν γίνει και για την ε, προσπάθεια εναρμονισμού που δημιουργεί ένα ε, δυσχερές πεδίο εφαρμογής και δυσκολίες εγγενείς σε αυτό το πεδίο. Είναι λοιπόν αυτό μια ολιστική βάση και προσέγγιση από πλευρά της προσέγγισης των κρατών μελών για ένα δικαιοδοτικό πλαίσιο ενιαίο και κοινό. Και κάθε φορά όταν προσπαθούμε να δράσουμε σε αυτό το πλαίσιο των επιμερισμένων αρμοδιοτήτων ανησυχούν σε σχέση με την ε, <clears throat> ε, η φαρπαγία στο αποκαλέσω έτσι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων τους. Δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε λοιπόν ευθύ εξ αρχής αυτή την πρόταση με μια πρόσθετη συνιστόσα. Και υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό επιχείρημα. Εργαζόμαστε για την ενιαία εσωτερική ψηφιακή αγορά. Και είχε ζητηθεί να προετοιμαστούν κανόνες και κανονισμοί για τις συναλλαγές ε, ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, πράγμα το οποίο κάναμε. Ευθύς εξ αρχής είχαμε ένα ανοιχτό πνεύμα και πλαίσιο σε σχέση με την, τον επιμερισμό αυτών των κανόνων για το διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου ότι δεν είναι ιδανικός και ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα. Και θα επιταχύναμε το έργο της επικαιροποίηση και εξυγχρονισμού ώστε με την οδηγία για τις εγγυήσει να μπορέσουμε ταχύτατα να συλλέξουμε τα αναγκαία αξιόπιστα στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πώς θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια κοινή παρόμοια προσέγγιση με στοχοθέτηση για συμβατικούς κανόνες offline στις συναλλαγές, ώστε ένα ενιαίο, σε ένα ενιαίο πλαίσιο να μπορούσαν να εφαρμοστούν. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Επιταχύνουμε σε σημαντικό βαθμό το έργο το οποίο επιτελούμε σε αυτή την πρώτη φάση όπως την προσεγγίζουμε για το εγχείρημα refit έχουμε έξι οδηγίες που πρέπει να καλυφθούν. Είναι επιπλέον την πρόσθετη αξία σε σχέση με τα δικαιώματα καταναλωτών, σε σχέση με τις πρόσφατες διατάξεις που υιοθετήθηκαν ε, πρόσφατα. Πρέπει λοιπόν μια συνολική επισκόπηση να διασφαλιστεί. Θα σας διατεθούν όπως προανέφερα αυτά τα στοιχεία κατά τον μήνα Ιούλιο. Τον Σεπτέμβριο και αναλαμβάνω αυτή την δέσμευση εδώ και σήμερα ενώπιόν σας, θα υπάρξει παγιοποιημένη, πάγια έκθεση <clears throat> και κατά πόσον είναι, <clears throat> μπορεί να ε, συστηθεί ή όχι, αυτά τα στοιχεία του refit να μπορέσουν να ενταχθούν και να τροφοδοτήσουν την πρόταση για τις ε, συμβατικές πράξεις, ε, για τις πράξεις ψηφιακού περιεχομένου. Θα συλλέξουμε τα στοιχεία και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τον εναρμονισμό offline. Εφόσον θα έχει διασφαλιστεί πιο πριν ότι αυτό θα είναι εφικτό, θα είναι βιώσιμο και θα έχει και μια πρόπτικη να εγκριθεί στο μέλλον και από το Συμβούλιο. Και τότε θα προσέλθουμε σε, σε εμάς στο Ευρωκοινοβούλιο με αυτή την πρότασή μας για μια τέτοια οδηγία για να συνεξετάσουμε τη δυνατότητα να προσθεθεί αυτή η συνιστόσα των κανόνων του παιχνιδιού offline στο κοινό πλαίσιο. Έχω διαπιστώσει και ανοιχνεύσει το κατεπήγον του χαρακτήρα, όχι μόνο από πλευρά σας, αλλά και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό θέλουμε αυτά τα στοιχεία να τα, να τα έχουμε στη διάθεσή μας το δυνατόν ταχύτερα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε σχέση με τις δράσεις μας αυτή την προσπάθεια. Το refit όμως θα ακολουθήσει σύντομα εν ευθέτω χρόνο μετά από αυτή την πρώτη προσέγγιση. Θα επανέλθουμε σε σας λίγο αργότερα, ε, μεταγενέστερα. Αυτά ήθελα να σας πω και για να γνωρίζετε το εύρος για τις ερωτήσεις που έγιναν για το refit. Έχουμε έξι οδηγίες ε, υπό το refit όπως προανέφερα. Η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές, ε, για τις εγγυήσεις, για τους όρους συναλλαγών, για τις τιμές και για την οδηγία για τις διαφημίσεις και για τις επιπτώσεις. Για να απαντήσω στην κυρία Χαράσοβα ότι άκουσε λέει ψιθύρους ότι θα υποβάλαμε μια πρόταση σχετικά. Άκουσα πολλούς ψιθύρους αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κανέναν από αυτούς τους ψιθύρους. Αρκετοί επίτροποι εξετάζουν τις δυνατότητες του B2B και υπάρχουν μελέτες ε, υπό εκπόνηση. Μπορεί να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα υστερότερα. Δεν μπορώ τώρα να δεσμευθώ και να δώσω στοιχεία αν θα γίνει εφέτωση του χρόνου αυτό. Αυτό που κάνουμε σε σχέση με την προστασία καταναλωτών και για τα ψηφιακά επικεντρώνεται απόλυτα στις σχέσεις B2C. Για το θέμα της ε, αφαιρεγγιότητας επικεντρωνόμαστε σε σχέση με την ε, ενότητα αγοράς, την Ένωση Αγορών, επ' αυτού και οι υπηρεσίες μου εξετάζουν τα, τις δυνατότητες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προανέφερε ο κύριος Σβάμπ, ότι υπάρχουν πολλά άτομα που λόγω του, της κατάστασης έχουν ε, συνάψει ε, δάνεια τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και απέβησαν εις βάρος τους. Ε, πρέπει να αναζητηθούν λύσεις τώρα σε άλλα θέματα αφαιρεγγιότητας που οδηγούν πολλές φορές σε πραγματικές τραγωδίες, ατομικές τραγωδίες που υφίστανται πολίτες. Πρέπει να δούμε το θέμα σε σχέση με την εμπορική προσέγγιση, γιατί με την εμπορική αφαιρεγγιότητα μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιακών Αγορών Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους δυσχέρειες με ε, έγκαιρη αναγνώριση ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων και δυνατότητες αναδιάρθρωσης των δανείων αυτών ώστε να μπορέσει κάτι να γίνει για τους ανθρώπους αυτούς. Το αποκαλούμε ε, πρόταση insolvency για την μη ρευστότητα ή αφαιρεγγιότητα και πρέπει να δούμε και σε σχέση με τα κράτη-μέλη θέλουμε να εισαχθούν κοινοί κανόνες ε, για την ε, εμπορική ε, χρεοκοπία ή μη εξυπηρέτηση δανείων και την ατομική μη ικανότητα εξυπηρέτησης δανείων και αφαιρεγγιότητα. Για μένα προσωπικά εγώ θα προτιμούσα να υποβάλαμε μια πρόταση για την αηφορία του επιχειρήν την αηφορία σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Αν, όπως για παράδειγμα στις ΕΠΑ ακολουθεί το μια διαφορετική προσέγγιση θα μπορούσαν να βοηθηθούν επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι ε, κλείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα ε, φλέγον θέμα. Πρέπει να επιταχύνω, το γνωρίζω, προστασία δεδομένων υπό το φως όλων αυτών των απολύσεων στο διαδίκτυο και την ε, δυνατότητα προστασίας των δεδομένων. Γνωρίζετε ότι είναι διτό αυτό σε σχέση με τις δικές μου αρμοδιότητες επί των ε, χαρτοφυλακίων αυτών. Πρέπει να παραμείνουμε συνεκτικοί και με συνάφεια στους κανόνες όσον αφορά τις ε, προοπτικές και δυνατότητες για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί πρέπει να εγκριθούν υπό το πλαίσιο της προστασίας ε, των δεδομένων μέχρι τον Μάιο 2018 πιο πριν θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός, πριν από την, ε, τον καθορισμό των νέων κανονισμών μας. Τι θέλω να πω, δεν ολοκληρώνεται το έργο, ούτε ολοκληρώθηκε με αυτό, μόνο ξεκίνησε με αυτό το εναρκτήριο λάκτισμα. Τρία πράγματα πρέπει να πετύχουμε. Να δημιουργηθεί μια ενιοποιημένη, ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή αφήνει πολλές διακριτικές εξουσίες όσον αφορά τις κυρώσεις ε, ε, ο κανονισμός αυτός, σε σχέση ε, με τα περιθώρια που δημιουργούνται και πρέπει να δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό που είναι σημαντικό για τους καταναλωτές και θέλω να το τονίσω είναι του χρόνου το 2017 θα γίνει μια πολύ μεγάλων διαστάσεων εκστρατεία ώστε να μάθουν, να γνωρίσουν οι καταναλωτές και να εξοικειωθούν με τα δικαιώματα που έχουν στην Ευρώπη ώστε να μπορέσουν την ιδιωτική τους σφαίρα, την ιδιωτική τους ζωή να την προστατέψουν με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Διότι οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιούν τους κινδύνους ε, που υφίστανται μέσα στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα και πρέπει έχοντας συνειδητοποιήσει αυτούς τους κινδύνους να γνωρίζουν τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν και θα διεξαχθεί μια πραγματικά έντονη μεγάλη σε εκστρατεία. Θέλουμε και στην νομοθεσία όπως στις ρυθμίσει για την προστασία δεδομένων συνεπιπρόσθετα την ε, διατήρηση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών. Με αυτή την εκστρατεία θέλουμε να διασφαλίσουμε την φιλοσοφική αρχή ότι πρέπει οι πολίτες να είναι κυρίαρχοι, να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα στα προσωπικά τους δεδομένα. Στα δεδομένα του συνολικά. Αυτό αφορά και την πρόταση για τις ψηφιακές συναλλαγές και συμβάσεις. Να ενημερώνονται οι πολίτες πώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον θα χρησιμοποιηθούν και θα διατεθούν. Πρέπει να έχουν, να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν αυτά τα δικαιώματα. Αν ανακοπεί η σύμβαση, η συμβατική σχέση πρέπει αμέσως να μπορεί να ανακοπεί, να διακοπεί και η χρήση δεδομένων από οποιουσδήποτε αυτών των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Μας κάνετε δηλώσεις ε, ε, πολλές. Ε, αυτό σημαίνει ότι εσείς ζητάτε ας πούμε πίσω τα στοιχεία για, τα, για τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχετε το κάθε κλικ που γίνεται. Τι, τι, γίνεται, δηλαδή πώς γίνεται όταν χρησιμοποιούνται μεγάλοι αλγόριθμοι για, για τα big data γιατί ακούμε από τις σχετικές εταιρείες και, αυτοί, αυτούς που δουλεύουν με την ε, ε, οικονομία του μοιράσματος, τη sharing economy, ότι ε, αυτά είναι προβληματικά πράγματα. Δηλαδή προσπαθούμε να, κάνουμε μια, να νομοθετήσουμε από τη μία πλευρά και δημιουργούνται προβλήματα από την άλλη. Εμείς θέλουμε πραγματική ψηφιακή οικονομία και θέλουμε πραγματικά σωστή και λειτουργούσα νομοθεσία. Ωραία. Και να σιγουρευτούμε ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν και οι άλλοι. Ε, ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει επιστρέφω τα στοιχεία, αλλά πάντως ε, το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει πάυση της δυνατότητας χρήσης των στοιχείων και οπωσδήποτε θα ενδυναμωθούν τα δικαιώματα των, ε, ανθρώπων, των ατόμων από τη στιγμή που θα τους δοθούν νέα δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα την προστασία, ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ενισχυθούν οι διαδικασίες επί παραβάσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται στοιχεία ή ψηφιακά περιεχόμενα. Ε, με σοκάρισε η συχνότητα πούμε ε, τέτοιων παραβάσεων κυρίως σε περιπτώσεις ποδοσφαιρικών αγώνων όπου 85% χρησιμοποιούνται τα ιδιωτικά ε, στοιχεία των ε, ατόμων. Και επομένως, ναι, θέλουμε να ε, επιφέρουμε τα απαραίτητα εχέγγυα, τα απαραίτητα όσον αφορά τους αλγόριθμους είμαστε ε, σε διαρκή επαφή ε, με τους παρόχους ε, IT στον τομέα της ασφάλειας. Και επιμένω ιδιαίτερος ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι αυτοί. Όταν προσπαθεί κάποιος να βρει την, ε, το, το παράνομο ε, ε, την, αυτή την φάση της παρανομίας τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ανακόπτεται η πρόσβασή του στο περιεχόμενο και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και σε συνεργασία και σε διάλογο με τους παρόχους τεχνολογίας IT. και η συζήτηση βεβαίως θα πρέπει να γίνει ε, στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτή. Τώρα, πώς μπορέσουμε να ε, τους σταματήσουμε να χρησιμοποιούν τους αλγόριθμους αυτούς ε, για εμπορικούς σκοπούς, δεν γνωρίζω αλλά πάντως η βούλησή μας κατά της πρακτικής αυτής είναι σαφής. Ωστόσο είναι ένα, ένας τομέας ο οποίος αναπτύσσεται ταχύτατα και επομένως θα ξανα κάνουμε τη συζήτηση σχετικά με το πού μέχρι πόσο μπορούμε να φτάσουμε. Η κυρία Κοράτσα το είπε προηγουμένως, δεν θα πρέπει να κάνουμε υπερβολική ε, νομοθέτηση, over-regulation. Ε, ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και οπωσδήποτε τα μέτρα μας να είναι σωστά και αναλογικά. Αλλά αυτό το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί οπωσδήποτε περαιτέρω. Όσον αφορά την ε, οικονομία του μοιράσματο, αυτή τη sharing economy, είναι στην ουσία ε, υπηρεσίες που παρέχονται από καταναλωτή σε καταναλωτή. Θέλουμε εδώ ε, ε, ε, να προστατεύσουμε τους εμπορευόμενους, θέλουμε να εξηγήσουμε πώς θα εφαρμόζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού όταν προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Όσον αφορά τις μονοπρόσωπες εταιρείε. Δεν έχουν μείνει και πολλά μετά από τις διαπραγματεύσεις. Επιμένω, είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στον 21ο αιώνα και επομένως θα πρέπει να είναι εύκολη η επιγραμμική ε, εκκίνηση μιας ε, εταιρείας ειδικά μιας μονοπρόσωπης ε, εταιρείας ε, με ένα ευρώ ας πούμε κεφάλαιο για την ίδρυση της εταιρείας. Ε. Θυμάμαι πόσο δύσκολα ξεκίνησα την επαγγελματική μου ζωή και ή αναγκάστηκα να πληρώσω πολλές χιλιάδες τσεχικές κορώνες που ήταν πολλά χρήματα για να μπορέσω να ξεκινήσω την ε, επαγγελματική μου δραστηριότητα. Θέλω λοιπόν να δώσω ευκαιρία στους ανθρώπους που ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Αλλά τώρα ε, ε, υπάρχουν πολλές, πολλά και σοβαρά εχέγγυα πολλές προστατευτικές δικλίδες για τους εργαζόμενους ε, για το κοινό που θα πρέπει να ξέρει ε, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ε, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαδικασία ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για την ίδρυση μιας τέτοιας εταιρείας. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερος προσφυλές και θέλω να το προωθήσω. Κίνα και ασφάλεια προϊόντων. Το Σάββατο πάω στην Κίνα και την Δευτέρα θα ξεκινήσουμε τις ε, συζητήσεις. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν θέλουμε ε, τα προϊόντα τους. Εγώ έχω ε, μιλήσει επανειλημμένως και με την ε, Αμερικανίδα Υπουργό Εμπορίου ε, και έχουμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε από τις κινέζικες αρχές μεγαλύτερο έλεγχο όλων των εμπορευμάτων που προορίζονται για την αμερικανική ή την ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι 60 με 62% των ανιχνευθέντων ως επικινδύνων ε, ε, αγαθών ε, να προέρχονται από την Κίνα. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, θέλω να επανέλθω από την Κίνα με συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα. Αυτό, ε, σε αυτό προσβλέπω. Μήπως, λέει η Πρόεδρος, να αρχίσουμε με τον επόμενο κύκλο των ερωτήσεων. Η κυρία Γραπίνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύρια Επίτροπε. Καταρχήν ευχαριστώ που προσήλθατε, κυρία Επίτροπε, και μπορούμε να διεξαγάγουμε αυτή τη συζήτηση. Παρακολούθησα τα πάντα με μεγάλη προσοχή, όλα όσα είπατε και αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Γι' αυτό τρία σημεία μόνο επιλέγω, σε αυτά τα θα επικεντρωθώ. Καταρχήν πρώτα είναι σημαντικό οι καταναλωτές και τα νομικά πρόσωπα να μπορέσουν να καλυφθούν, όχι μόνο τα φυσικά άτομα. Και τα οι, οι νομικές οντότητες είναι σημαντικές ε, και αυτές ε, όσον αφορά τις πρώτες ύλες, ε, την επεξεργασία τους και οι τράπεζες, τραπεζικά ιδρύματα. Πολλές φορές υπάρχουν δυσκολίες λόγω των αθέμητων εμπορικών πρακτικών που αναφέρθηκαν ως πρόβλημα. Όσον αφορά τις τράπεζες, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν και τα θέματα καταναλωτών να εξεταστούν και σε αυτό το πλαίσιο. Και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου πρέπει να καλύπτονται. Ερώτηση, τι θα κάνετε, Στοχεύεται να πράξετε ώστε να μειωθεί, να απαμβληθεί η πίεση, ιδιαίτερα όσον αφορά την πίεση που δημιουργείται από μονοπόλια και με το θέμα του εναρμονισμού προς όφελος των καταναλωτών. Τι μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, για, για πρακτορία τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γραφεία τουρισμού, όταν υπάρχει, για παράδειγμα, έγινε μια ε, διασυνοριακή συνάντηση ε, στη Σερβία, όταν φυσικά πρόσωπα που είχαν αγοράσει υπηρεσίες ε, τουριστικές είχαν φέρει με λεωφορεία είχαν μεταφερθεί και είχαν μεταφέρει αντικείμενα και εδώ ακριβώς και σε σχέση με την ε, ε, γλώσσα που ε, ε δεν αναφερόταν υποχρεωτικά στη χώρα προέλευσης η γλωσσική αυτή θα έλεγα ε, εναρμονισμένη ρύθμιση και για λεωφορεία, πούλμαν και για τις οδηγίες χρήσεως αυτών αντικειμένων και των οχημάτων αυτών. Πρέπει να εναρμονιστούν όλα αυτά τα πλαίσια και το πλαίσιο ασφάλειας προϊόντων. Επί 25 χρόνια εργάστηκα σε σχέση με την παραγωγή και είχα ε, συσχετιστεί και με προϊόντα που εισήγονται από την Κίνα. Εδώ είναι σημαντικό όχι μόνο να έχουμε απαγορεύσει σε σχέση με κάποια χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εισαγόμενα εμπορεύματα, αλλά να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την ίδια την Ευρώπη. Νομικά πρόσωπα ε, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ευρώπη. Ποιοι έλεγχοι μπορούν να επιβάλλονται λοιπόν σε σχέση με τέτοια προϊόντα προέλευσης Κίνας. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τους ε, ε, ελέγχους εξαγωγών από τους Κινέζους, πρόκειται και για τους ελέγχους εισαγωγών από εμάς τους Ευρωπαίους εδώ άμεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι εν μέρει απαντήσατε στα ερωτήματά μου, αλλά θέλω να επισημάνω κάποια θέματα. Οι δύο προτάσεις, ε, πωλήσει online και offline για ψηφιακά προϊόντα, ε, ήδη βρίσκονται στη διαδικασία τη δική μας. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τα δεδομένα που αφορούν στον καταναλωτή. Βεβαίως δεν έχουμε ιδέα το πώς θα τα πειράσει όλα αυτά το refit. Επίσης, συμφωνώ με την Εβελίν ότι οι δύο προτάσεις δημιουργούν σύγχυση στους ε, καταναλωτές. Κυρίως γιατί υπάρχουν κάποια οριακά προϊόντα όπως ε, χειροπιαστά με ψηφιακό λογισμικό που δεν είναι εύκολο να ταξινομηθούν με βάση αυτές τις ε, προτάσεις. Μήπως μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς όλο αυτό το refit θα επηρεάσει την σα για τον καταναλωτή και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να συνδυάσει τις ε, δύο αυτές ε, προτάσεις με το refit. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριο Στέφανετς, κυρία Επίτροπε, ε, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή για την τυποποίηση, την απλούστευση για τους ανθρώπους που θέλουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο να προτίθεστε επίσης ε, να προτείνετε και άλλου είδους απλουστεύσεις για διαφορετικές ε, επιχειρήσεις για μονοπρόσωπες εταιρείες, παραδείγματος χάρη Σα ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Κυρία Επίτροπε, υπάρχει μια πρόταση την οποία αναμείναμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Η βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Σημαντική προϋπόθεση και όρος για την κοινή ψηφιακή εσωτερική αγορά. Δεν θα πρέπει όμως αποκλειστικά να επικεντρωνόμαστε στο διαδικτυακό εμπόριο. Και με ενδιαφέρει επίσης να δούμε τις προτάσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα οδηγία όσον αφορά την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Τι είναι εκείνο το οποίο σχεδιάζετε και έχετε προγραμματίσει από πλευρά σας, διότι υπάρχει ένας κανόνας που προβλέπει ότι θα πρέπει να επιτυγχάνεται ποσόστοση δύο τρίτων και όχι μόνο ενός ημίσεως. Αυτό είναι πολύ υψηλή προϋπόθεση. Θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και πιστεύω ότι δεν πρέπει να δίνουμε δυνατότητα να παρακάμπτονται ε, διατάξεις ε, ε, κατά του αθέμητου, των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Σημαντικό είναι τα όργανα, τα κρατικά όργανα και οι κρατικές αρχές σε περιφερειακό επίπεδο να μπορούν να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά και είναι σημαντικό να ανταλλάσσονται πληροφορίες και στοιχεία αν υπάρχει κάποια υποψία αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και επιπλέον θεωρώ ότι και διμερός διμερείς επαφής, επαφές μπορούν να είναι σημαντικές και ελπίζω ότι θα ληφθεί αυτό πλήρως υπόψη για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. And the last one is Thank you. Τελευταία η κυρία Γιακονσάρη. Ε, κυρία Γιακονσάρη, πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι αυτό μετατίθεται, μετακινείται και γίνεται μια εργαλειοθήκη IT είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια αυτό το θέμα στην ε, κοινωνική μας πολιτική, στις πολιτικές μας. Να το συζητήσουμε ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες περί πρόκειται υποστηρίζει την πρόταση της ΙΝΚΟ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αλγόριθμοι θα πρέπει να αποτελέσουν ένα προ, πρόγραμμα πιλωτικό ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποια θέματα θα πρέπει πολιτικά να καλυφθούν και να ρυθμιστούν ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται για τη χρήση τέτοιων στοιχείων. That's είναι οι ερωτήσεις μας υπενθύμησαν ότι πριν από δυόμιση χρόνια δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να καλυφθούν θέματα ε, καταναλωτών από την Επιτροπή και δείτε που φτάσαμε σήμερα. Η κυρία Γιούροβα για το θέμα για τα νομικά πρόσωπα ήδη προηγούμενα είπα B2B σχέσεις είναι εκείνες ε, που εξετάζονται αυτή τη στιγμή στις μελέτες που βρίσκονται υπό εξέλιξη και στο refit και την επικαιροποίηση και εξυγχρονισμό. Και ουσιαστικά το βασικό στοιχείο στην πολιτική προστασίας καταναλωτών είναι η προστασία του πιο αδύναμου κρίκου. Και προφανώς βλέπουμε ότι στο συσχετισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των τεράτων των τεραστίων πελωρίων επιχειρήσεων υπάρχει μια μη ισορροπή σχέση. Είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να υπάρξει ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας, ε, πράγμα το οποίο ε, βέβαια ε, εν σπέρματι εν υπάρχει στην νομοθεσία μας, αλλά πρέπει πιο συγκεκριμένα να δούμε πώς θα μπορέσει να καλυφθεί σε σχέση με τα μετεξελισσόμενα και νεοαναφιόμενα προβλήματα που διαρκώς ε, ε, ε, αναφύονται και πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά θα τα ρυθμίσουμε και όπως είπα αυτό μπορεί να ακολουθήσει και ιστερότερα. Τώρα συγκεκριμένα για δυνατότητες συγκεκριμένης προστασίας. Συμφωνώ απόλυτα ότι οδηγίες στα αγγλικά ή σε μια άλλη γλώσσα δημιουργεί μια συμμετρία πληροφόρησης που δεν θα πρέπει να την ανεχόμαστε. Ε, πρέπει με συγκεκριμένα παραδείγματα να αντιμετωπιστεί αυτό, διότι είναι θέμα εθνικών ρυθμιστικών αρχών, εθνικών οργάνων που πρέπει να παρεμβαίνουν προς ρύθμισή τους. Και πρέπει επίσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο να μπορέσουμε πανενοσιακά να δράσουμε. Και σε, με συγκεκριμένες ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις και δράσεις θα μπορούσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Πώς θα μπορούσε τώρα η προστασία δεδομένων, η κυρία Μπόρζαν το θέμα αυτό το ανέφερε, να διαμορφωθεί. Όπως είπα, είμαστε αρμόδιοι και για την προστασία καταναλωτών και για την προστασία των δεδομένων. Όλα όσα θα πράξουμε υπό το refit στην ε, κλίμακα αυτή των πρωτοβουλειών μας θα πρέπει να είναι συμβατά και να συνάδουν με την προστασία δεδομένων και πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο, διότι έχουμε υπηρεσίες που εργάζονται μέσα στο πλαίσιο της Επιτροπής προς τη μία και άλλη κατεύθυνση και πρέπει με έναν συνεκτικό τρόπο να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί βρείτε κάποιο συγκεκριμένο εξειδικευμένο πρόβλημα για την προστασία δεδομένων, να μου το γνωστοποιήσετε άμεσα διότι πραγματικά θα ήταν μεγάλο λύστημα, θα ήταν παράπτωμα αν δεν μπορούσαμε να δράσουμε ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για την προστασία δεδομένων όπως και με άλλες νομοθετικές δράσεις μας. Τώρα, πράγματι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε είναι εργαζόμαστε για τη δέσμη μέτρων για τη νέα νομοθεσία για την ψηφιοποίηση όσον αφορά την ε, νομοθεσία για τις επιχειρήσεις. Δεν έχει πάρει ακόμα συγκεκριμένη τελεσίδικα μορφή. Έχουμε μια ομάδα πραγματογνωμόνων που ε, μας συμβουλεύει για τις αλλαγές όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο και την ψηφιοποίηση. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο αφετέρου πρέπει να δούμε ότι ε, συνεπάγονται και κάποιους κινδύνους που πρέπει να καλυφθούν. Αυτά εξετάζουμε τώρα σε σχέση με την, το πλαίσιο της οδηγίας και των δρασεών μας. Θα υποβάλουμε πρόταση του χρόνου το 2017 σε σχέση με τη μετεξέλιξη του εταιρικού δικαίου και θα αναλώσουμε περισσότερο χρόνο σε σχέση με τα θέματα επιχειρήσεων και τα ψηφιακά. Ναι, κύριε Φόρτ, το γνωρίζω ότι οι αλγόριθμοι δεν αφορούν ε, ε, αποκλειστικά και μόνο θέματα ε, μ, αναζωπήρωσης ε, μίσους ή λόγων και κηρυγμάτων μίσους. Θα πρέπει να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πλαίσιο διαλόγου με τις, τους εμπλεκόμενους και τις επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις IT, ώστε να μπορέσουμε να εισαγάγουμε και να πράξουμε νομοθεσία για αυτές τις ε, ε, ε, δυνατότητες. Με τους αλγόριθμους τι μπορεί να γίνει. Μόνο αν υπάρχει παραβίαση ή παράβαση νομοθεσίας προστασίας δεδομένων μπορεί να αναλυφθεί κάποια πρωτοβουλία. Ή αν συνεπάγονται κάποια παραπλανητική πολιτική εξαπάτησης που τότε μπορούμε να εμπλακούμε και να προσπαθήσουμε να κυρώσουμε. Συνεχίζω στη γλώσσα μου προς την ε, Ευρωβουλευτή ε, που ομιλεί τη γλώσσα μου. Ε, τώρα, αν όλα αυτά θα επαρκέσουν, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει το μεγαλύτερο ποσοστό των ε, πολιτών μας ε, να καλύφθει ε, τέσσερις φορές ετήσια όταν για παράδειγμα υπάρχουν τέσσερις φορές παρα, τέσσερις παραβιάσεις ή παραβάσεις ανά έτος. Κάνουμε λόγο για ένα ευρύτατο πεδίο εδώ και γι' αυτό θα ήθελα να μπορέσουμε να εγκρίνουμε το δυνατόν νωρίτερα την οδηγία για την συνεργασία σε σχέση με την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Έτσι οι ενώσεις, οι σύλλογοι προστασίας καταναλωτών και εθνικές αρχές θα μπορέσουν να συνενώσουν δυνάμεις ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω αυτά είναι όλα όσα ήθελα να αναφέρω. Αν ξέχασα κάτι να μου το αναφέρετε να επανέλθω. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες της Επιτροπής μας για σήμερα το πρωί. Θα ξανασυναντηθούμε στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας.